Καλημέρα σας. Λοιπόν για την καθυστέρηση, αλλά περιμένουμε και άλλους συναδέλφους που είναι λιγότερο συνεπείς από εμά, αλλά σήμερα ο χρόνος μας είναι μετρημένος και από αυρότητα προς τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μοχαμέτ Σαλέμερ Σαλέκ. Καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Όπως γνωρίζετε το πρώτο σημείο είναι η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα με συγκεκριμένη αναφορά στα γεγονότα τα οποία συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Σε αυτή τη συζήτηση συμμετέχει και η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Μαγκρέμπ που εκπροσωπείται από τον πρόεδρο Παντζέρη, τον οποίο χαιρετίζω. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον εκπρόσωπο του μετόπου Πολυσάριο, τον υπεύθυνο για τις εξωτερικές σχέσεις. Ξέρετε ότι και υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου θα πάρει το λόγο, αλλά σε μια συνάντηση που θα ακολουθήσει ανάμεσα στις 11 και 11 και Ο κύριο είναι χαρά για μας που είχατε τη δυνατότητα να είστε εδώ σήμερα και να έρθετε σε επαφή με τους συναδέλφους. Όπως γνωρίζετε το Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα υιοθέτησε ένα ψήφισμα για την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα και εκεί εκφράζονται ορισμένες εκτιμήσεις για το πρόβλημα και είναι φυσικά σωστό να μπορέσουμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις στην Δυτική Σαχάρα και έτσι να επιτρέψουμε σε όλους τους εμπλεκομένους, Μαρόκο, την δική σας οργάνωση και τους συναδέλφους να ανταλλάξουν απόψεις. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ξέρω ότι έχουμε ήδη συναντηθεί βέβαια και είστε αποτελεσματικός στην επικοινωνία και στα δέκα λεπτά τα οποία σας έχουμε δώσει. Ελπίζω να τα σεβαστείτε και να παρουσιάσετε με πλήρη τρόπο το θέμα που έχουμε όλοι μπροστά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλή σας μέρα. Θα κάνω την ομιλία μου στα Ισπανικά, γιατί έχω και τη μετάφραση στα Αγγλικά, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω τον αρμόδιο που θα τη μοιράσει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έρχομαι εδώ μετά την πιο σημαντική που έχουμε ζήσει μετά την κατάπαυση του πυρός του 1991 μεταξύ του με το και του Μαρόκου και μια στιγμή μάλιστα που τα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας, τα κατεχόμενα από το Μαρόκο, ζουν ε, σε ένα κλίμα εκφοβισμού μετά την υιοθέτηση των ε, πιο δρακόντιων ε, μέτρων που έχει εφαρμόσει μέχρι στιγμής ε, η μαροκινή κυβέρνηση εις βάρος του λαού της Δυτικής Σαχάρας και της πρωτεύουσας Λαγιούν. Έρχομαι παρόλα αυτά ενώπιόν σας με μία ελπίδα. Με την ελπίδα ότι τα πρόσφατα επεισόδια της Δυτικής Σαχάρας θα σηματοδοτήσουν μια κρίσιμη στιγμή, μια αποφασιστική στιγμή για το λαό μου και την έναρξη μιας σοβαρής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ μιας δημοκρατικής λύσης στη Δυτική Σαχάρα. Μιας λύσης που θα επιτρέψει στο σαχαροίτικο λαό να επιλέξει το πεπρωμένο του. Μια διαδικασία αυτοδιάθεσης θέλουμε για το λαό μας. Κάτι αντίστοιχο συνέβη στην Αμμύμπια. Νομίζω ότι το δικαίωμα μας αυτό είναι δικαίωμα που συνάδει με το Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς, γιατί γνωρίζετε τα γεγονότα. Η Δυτική Σαχάρα είναι η τελευταία απικία της Αφρικής. Και από το 1963 βρίσκεται στον κατάλογο του ΟΗΕ ως μια αυτόνομη περιοχή. Και μετά την απόφαση της Ισπανίας να εγκαταλείψει την περιοχή το, το 1975, το Διεθνές Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απουσία οποιονδήποτε διεκδικήσεων ή νομικού συνδέσμου που θα ακύρωναν τη διαδικασία αυτοδιάθεσης του Σαχαροϊτικού λαού που θα έπρεπε να εκφραστεί με λαϊκή τιμιγορία. Το δικαστήριο ρητά απέρριψε τις ε, διεκδικήσεις και αξιώσεις του Μαρόκου επί της ε, επικράτειας της Δυτικής Σαχάρας. Το 1991 το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ένα σχέδιο που προβλέπει κατάπαυση του πυρός και, αυτοδιάθεση, ε, και δημοψήφισμα για αυτοδιάθεση στη Δυτική Σαχάρα που έπρεπε να έχει γίνει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το 1992. Έχουν περάσει όμως 20 χρόνια και δεν έχει διοργανωθεί αυτό το δημοψήφισμα παρόλο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Μετόπου και του Μαρόκο. Το Μαρόκο εμπόδισε τη διεξαγωγή αυτού του δημοψηφίσματος. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή δεν είναι ο εντοπισμός των ψηφοφόρων επιχείρημα του Μαρόκου. Αλλά, όπως είπε ο κ. James Baker, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος φοβόταν το Μαρόκο. Σε μια συνέντευξη ο κ. James Baker, ο πρώην ειδικός εντεταλμένος στο ΙΕ στη Δυτική Σαχάρα, είχε πει ακριβώς αυτό. Ότι όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στο δημοψήφισμα, τόσο πιο ε, μεγαλύτερο εκνευρισμό έδειχναν οι Μαροκινοί απέναντι στην πιθανότητα να χάσουν το δημοψήφισμα. Το Μαρόκο προτιμά να κερδίσει χρόνο ελπίζοντας ότι η διεθνή κοινότητα θα δεχθεί αυτή την παράνομη κατοχή. Όπως έδειξε όμως η τραγωδία του Λαϊγιούν, Κανείς δεν είναι υπέρ της παράνομης κατοχής αυτής από το Μαρόκο. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα του κόσμου που αναγνωρίζει τη μαροκινή κυριαρχία επί της Δυτικής Σαχάρας. Κανένας δεν αναγνωρίζει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, η δημοκρατία της ε, Σαχάρας είναι ιδρυτικό μέλος και πλήρες μέλος της ε, Αφρικανικής Ένωσης. Κάτι που δεν ισχύει για το Μαρόκο. Κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα της 25 ε, ης Νοεμβρίου για την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα έδειξε για μία ακόμη φορά το ρόλο του ως δημοκρατική συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να ζητήσουμε από αυτό το δημοκρατικό θεσμό που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκαινιάσει ένα νέο κεφάλαιο που μετά από 35 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσε να δώσει τα θεμέλια για ένα ειρηνικό, ασφαλές ε, και ευήμερο Μαγκρέπ που είναι γείτονα της Ευρω... Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δημοψήφισμα είναι το πρώτο βήμα για να πραγματοποιήσουμε αυτό το όραμα. Μια υπόσχεση άλλωστε που είχε δοθεί πριν από 20 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι η σημερινή συνεδρία σχετίζεται και με την επιθυμία σας να δείτε τι έγινε στο στρατόπεδο μουζίκ και στην πόλη Λαγιούν στις αρχές του Νοεμβρίου και για ποιο λόγο. Θα ήθελα να ρίξω λίγο φως σε όλες αυτές τις απορίες και τα ερωτηματικά. Από τις αρχές του Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, πολλές οικογένειες σαχαροϊτικών οικογενειών άφησαν, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους ε, στα κατεχόμενα και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα Λαγιούν για να εγκατασταθούν σε ένα μεγάλο στρατόπεδο, σε ένα μεγάλο καταβλισμό στα περίχωρα της πρωτεύουσα Λαγιούν. Και ο λόγος αυτής της ειρηνικής διαμαρτυρίας οφειλόταν σε μια αίσθηση ματέωσης και απογοήτευσης καθώς και απόγνωσης που αισθάνονταν οι Σαχαραουίτες για την ε, δινή οικονομική κατάσταση, τις διακρίσεις και την πολιτική περιθωριοποίηση την οποία τους επέβαλε η μαροκινή κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τους Σαχαραουίτες ως ε, πολίτες ε, ούτε καν δεύτερης ε, κατηγορίας, ακόμη χειρότερα. Αυτή η συσσωρευμένη ματέωση και απόγνωση των τελευταίων δεκαετιών σε συνδυασμό με την απομάκρυνση από τις οικογένειές τους οδήγησαν σε αυτή τη διαμαρτυρία. Και πολλές εκθέσεις, καθώς και εναέρειες φωτογραφίες, έδειξαν ότι περίπου 8.000 σκηνές και 26 με 30.000 ε, Σαχαραουίτες βρίσκονται στα τέλη Οκτωβρίου σε αυτό το καταβλισμό στα περίχωρα της Λαγιούν. Οι ειρηνικές και μη βίες αυτές διαμαρτυρίες οδήγησαν σε αύξηση της παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων του Μαρόκου γύρω από τον καταβλισμό αυτό και μία αύξηση των, ε, των περιορισμών σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε αλλοδαπή παρουσία γύρω από τον καταβλισμό. Επίσης εμποδίστηκε η πρόσβαση στην ζώνη αυτή και της ε, ειρηνευτικής δύναμης παρά την εντολή και τις επίσημες συμφωνίες που είχαν συναυθεί μεταξύ Μαρόκου και ΟΗΕ μετά την δολοφονία, τον πυραβολισμό από τις μαροκινές δυνάμεις ενός νεαρού 14χρονου Σαχαραουίτη, του Νάτζο Μιλγκέρχη, και τον τραυματισμό άλλων πέντε εφήβων που μετέφεραν τρόφιμα στον καταβλισμό στις 24 Οκτωβρίου, τα δρακόντια μέτρα και οι περιορισμοί αυξήθηκαν. Και το Μαρόκο ανενδίαστα και ξεδιάντροπα ξεκίνησε την τον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων με το μέτωπο Πολυσάρι από την αιγίδα του ΟΗΕ, προκειμένου να διαλύσει τον καταβλισμό στις αρχές του Νοεμβρίου. Ήταν δύσκολο να λάβουμε αξιόπιστες πληροφορίες εξαιτία των σοβαρών περιορισμών που μας είχε επιβάλει η μαροκινή κυβέρνηση στη Λαγιούν και στα προάστια της. Όχι μόνο για τους ειδικού επεσταλμένου, αλλά και για τους πρέσβει και για τους ευρωβουλευτέ, και για τις ανθρωπιστικέ δυνάμεις και για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Κανένας δεν μπόρεσε να εισέλθει στην περιοχή αυτή και μάλιστα ο Βίλι Μάγερ απελάθηκε όπως πολλοί άλλοι ευρωβουλευτές από τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία και άλλες χώρες. Βέβαια, μια τέτοια κατάσταση είναι απολύτως απαράδεκτη και γελιοποιεί τη δήλωση του Μαρόκου ότι δεν έχει να κρύψει τίποτα. Πολλαπλές ε, εκθέσεις ε, καταγγέλουν τη χρήση ε, βίας από το Μαρόκο για την καταστολή αυτής της ειρηνικής διαμαρτυρίας και μάλιστα και όπλων και πυρός. Είχαμε πολλά θύματα και εκατοντάδες ε, τραυματίες και αγνοούμενους από την καταστολή του Μαρόκου. Μάλιστα, πρόσφατη έκθεση της Human Rights Watch που δημοσιεύθηκε στις 26 Νοεμβρίου αναφέρει πολλές ε, αποτρόπες καταγγελίες για βασανιστήρια και κακοποίηση εις βάρος των, των διαδηλωτών μετά την απόπειρα του Μαρόκου να διαλύσει τον καταβλισμό αυτό. Μάλιστα φοβόμαστε ότι είχαμε και μια δολοφονία. Και φαίνεται ότι ο σαχαροϊδικός λαός στη Λαγιούν υπόκειται τις επιθέσεις ε, του μαροκινού καθεστώτος που προσπαθεί να αποκρύψει τις φρικαλαιότητες αυτές ε, και τις βαναυσότητες του από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολλά χρόνια εγκατάλειψης έζησε ο λαός της ε, Σαχάρας, της Δυτικής Σαχάρας απέναντι στην βάναυση συμπεριφορά του Μαρόκου και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια ευθύνη με την ε, πρωτοκαθεδρία της ε, Ισπανίας και της Γαλλίας. Η Γαλλία υποστηρίζεται στο Μαρόκο και η, η Ισπανία πρώην ε, απεικιοκρατική δύναμη εμποδίζουν οποιαδήποτε σοβαρή επίλυση Τη διένεξη αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλα αυτά έχει στα χέρια της ε, την δυνατότητα να εγκαινιάσει ήδη από σήμερα μια άλλη στρατηγική, μια νέα στρατηγική απέναντι στη Δυτική Σαχάρα. Καταρχήν, ε, η αποτυχία επίση του Μαρόκου για να ε, εφαρμόσει την εντολή τη Μενούρσου που επιτρέπει την εξαγωγή δημοψηφίσματο στο λαό της Δυτικής Σαχάρας με επιλογή και της ανεξαρτησίας, όπως συμφώνησαν τα συμβαλόμενα μέρη και ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ψήφισμα του 1991. Δεύτερον, η αποτυχία κατάρριψης της ε, γαλλικής αντίστασης ε, και της υποστήριξης των Μαρόκο, προκειμένου να τηρηθούν περισσότερο τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δυτική Σαχάρα. Μέχρι στιγμής καμία ανθρωπιστική δύναμη, μάλλον δύναμη διατήρηση τη Ειρηνή ε, σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου στερείται τέτοιων δυνατοτήτων. Και μάλιστα η αποτυχία τη εξασφάλιση τη κυριαρχίας του σαχαριώτικου λαού στο, στο φυσικό πλούτο τη περιοχή του είναι πραγματικά παραβίαση του διεθνού δικαίου. Μάλιστα η Ελευτική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Μαρόκου με βάση την οποία ευρωπαϊκά ελευτικά σκάφη μπορούν να αλλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Δυτικής Σαχάρας είναι παράβαση των δικαιωμάτων του λαού της Δυτικής Σαχάρας. Και μάλιστα αν ανανεωθεί αυτή η συμφωνία που λύγει το Φεβράριο του 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενεργήσει ως θεματοφύλακας της, του νόμου και να γίνει συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέλαμε να επιμείνετε τα χωρικά έδρα της Δυτικής Σαχάρας να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, γιατί αυτός ο Ελευτικό πλούτος είναι κληρονομιά του λαού της Δυτικής Σαχάρας και το Μαρόκο δεν έχει καμία νομική βάση για να περιλαμβάνει δική μας επικράτεια σε δικές του συμφωνίες. Θα πρέπει να διαβουλεύεται το λαό της Δυτικής Σαχάρας γιατί έχουμε, εμείς θα πρέπει να έχουμε την κυριότητα και την κυριαρχία στους φυσικούς μας πόρους. Και μάλιστα, όπως είπαμε και στην επιστολή που στείλαμε στο Συμβούλιο ασφαλεία στον ΟΗΕ, μετά τις επιθέσεις ε, του Μαρόκου της 15 η Νοεμβρίου, έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια αποφασιστική στιγμή. Το status quo δεν είναι πια επιλογή. Θα πρέπει να αλλάξουν όλα από εδώ και πέρα. Και παρά τις πιέσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χάρη στο ψήφισμά του, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς το Μαρόκο και στον κόσμο για τις ανησυχίες σας ως προς το Δυτική Σαχάρα. Αυτή είναι όμως μόνο η απαρχή. Το επόμενο βήμα θα είναι μια πιο ευφύης ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στη Δυτική Σαχάρα που θα ανταποκρίνεται στην αφοσίωση και την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές δίκαιο και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Με μια τέτοια πολιτική θα επηρεάσει και τη θέση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην όλη διένεξη. Οποιαδήποτε πρόοδος ό,τι αφορά το καθεστώς του Μαρόκου θα πρέπει να γίνει υπό τον όρο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη χώρα αυτή και τη στήριση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για τη διαδικασία αυτοδιάθεση του σαχαροϊτικού λαού. Μία τέτοια νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα αναγνωρίζει μία δίκαιη λύση στην σύγκρουση της Δυτικής Σαχάρας. Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση για όλους, δηλαδή μια περιοχή σταθερή και ειρηνική, προκειμένου να έχουμε μια σίγουρη και ευήμερη μεσογειακή λεκάνη. Αυτή είναι η βούληση και του Σαχαραϊτικού λαού. Ελπίζω να δημιουργηθεί το δημοψήφισμα και να γίνει και ο Σαχαροίτικος λαός ένας επικοδομητικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία μιας πιο θετικής και μιας πάγιας περιφερειακής αρχιτεκτονικής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ και πάλι για τη σημαντική ευκαιρία που μας δώσατε να απευθύνουμε ομιλία στην Επιτροπή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις, απορίες ή να ακούσω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σας έφερα και τεκμηρίωση για την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ολτσαλέκ. Δύο λεπτά θα μιλήσει ο κύριος Αλαφάνκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον εκπρόσωπο του μετά από Πολυσάριο, του κυρίου Σαλέμ Ολτσαλέκ. Και όντως έχουμε Μία σύγκρουση που κρατά εδώ και 35 χρόνια και τα τελευταία επεισόδια πραγματικά καταστρατηγούν κατάφορα τη διεθνή νομιμότητα όπως φαίνεται και από τα πολλαπλά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις προς τον εκπρόσωπο του μετώπου Πολυσάρη, που αργότερα θα επαναλάβω και στον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου. Η πρώτη ερώτηση είναι, Πώς αξιολογείται το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητάει που μάλιστα οι μαροκινές αρχές ε, το χαρακτήρισαν ως άδικο, εσπευσμένο και μεροληπτικό. Η δική σας εκτίμηση για το ψήφισμα αυτό ποια είναι. Δεύτερον, από τις ε, ειδήσει και τις πληροφορίες στον τύπο γίνεται λόγος για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς είπατε ότι φοβάστε ότι έγινε και μακελιό. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε του μετά από να μου δώσετε πιο ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των αγνοωμένων, για τον αριθμό των κρατουμένων, των τραυματιών. των νεκρών, οτιδήποτε στοιχεία έχετε για τα τελευταία επεισόδια. ζητήσατε την ε, παράταση της ε, εντολής της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών και σε θέματα παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια, μια τέτοια απόφαση θα τη λάβει το Συμβούλιο Ασφαλείας το ε, Τι προοπτικές έχει αυτό το αίτημα που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψηφισμά του. Υπάρχει πιθανότητα να σε αυτό το αίτημα και τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή υπό την αιγίδα του ειδικού εντεταλμένου του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Ο κύριος Γιάννης, δύο λεπτά. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Μετώπου Πολυσάριο για την παρουσία τους εδώ και να τους ευχαριστήσω και για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκάλεσε τους εκπροσώπους του μετόπου Πολυσάριου εδώ για συζήτηση και για ενημέρωση, είναι αξιοσημείωτο γεγονός από την άποψη των κοινοβουλευτικών πρωτοβουλειών. Όπως είπε ο κύριος Αλαφράγκα, αυτή η διένεξη κρατά εδώ και 35 χρόνια. Μία τέτοια σύγκρουση λοιπόν δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με ψυχρότητα, με αδιαφορία. Θα πρέπει να διακρίνουμε το πραγματικό από το φανταστικό, την πραγματικότητα από τις φήμες. Και μάλιστα η δικτατορία του Φράνκο, που ήταν ήδη πολύ άρρωστος όταν έγινε η πράσινη πορεία που οργάνωσε ο βασιλέας Χασάν του Μαρόκου, οδήγησε στην απομάκρυνση της ε, Ισπανίας από τη Δυτική Σαχάρα, από την διοίκηση τη Δυτικής και τότε έχασε και η Ισπανία τη δυνατότητα οποιασδήποτε επιρροή ή οποιασδήποτε συμμετοχής σε μία απόφαση του Σαχαροϊτικού λαού για αυτοδιάθεση, παρόλο που ήμασταν υπέρ αυτής της ε, αναγνώριση. Και το μόνο που έκανε η Ισπανία και που μπορούσε να κάνει και όλες οι διαδοχικές δημοκρατικές κυβερνήσεις και η Σοσιαλιστική και του Λαϊκού Κόμματος ήταν να υποστηρίξουν τη διαδικασία από απεικιοποίησης ε, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Και αυτή είναι μια διαδικασία που θα συνεχίσει η Ισπανία. Ε, μένω σε μια έκφραση που είπατε ότι είμαστε υπέρ ενός ε, σταθερού, ειρηνικού και ευήμερου Μαγκρέπ. Φυσικά. Και αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η μοίρα του σαχαριτικού λαού. Και νομίζω ότι η Ισπανία είναι από τις χώρες που προσφέρουν μεγαλύτερη ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια στους Σαχαραουίτες. Η δεύτερη αρνητική επίπτωση, ολοκληρώνω πρόεδρε, μισό λεπτό ακόμη. Η δεύτερη αρνητική επίπτωση της σύγκρουση αυτής είναι μια στάθεια στο Μαγκρέμπ και μια αντιπαράθεση Μαρόκου-Αλγερίας. Γιατί η Αλγερία ουδέποτε δεν αναφέρεται σε αυτές τις συζητήσεις, παρόλο που είναι σημαντικός παράγοντας. Θα ήθελα να σας θα παρακαλέσω να τηρήσετε το χρόνο, γιατί έχουμε μετρημένα τα λεπτά εδώ. Ο κύριος Βάγκλ, για δύο λεπτά. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Ε, νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις απαραίτητες για να βρεθεί μια τελική λύση στο πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν οφείλεται στα γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν λίγες εβδομάδες αλλά είναι η αναγνώριση ενός εγγράφου το οποίο αναγνωρίζεται θα έλεγα από, όλα τα, από όλες τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν αγνοούμε την κατάσταση, δεν αποστρέφουμε το βλέμμα μας από το πρόβλημα. Βλέπουμε ότι τίθεται εδώ ένα θέμα άγνοιας της διεθνούς τάξης και του διεθνούς δικαίου και ένα έντονο θέμα παραβίανων δικαιωμάτων. Με εκπλήσουν οι ενέργειες του Μαρόκου Εκπλήσωμε επίσης και από τις αντιδράσεις του μαροκινού κοινού που διαμαρτυρήθηκε έντονα για το ψήφισμα το οποίο κυκλοφορήσαμε. Νομίζω ότι η αντίδραση δεν ήταν δημοκρατική και αυθόρμητη και νομίζω ότι ήταν κακό το ότι υπήρξαν και περίεργες δηλώσεις κατά του ψηφίσματος αυτού από πλευράς Ισπανών πολιτικών. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι μέσω του ψηφίσματος αυτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέστειλε ένα μήνυμα προς το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να εμπλακεί έτσι περαιτέρω στην προσπάθεια αναζήτηση λύση στη Δυτική Σαχάρα, έτσι ώστε οι Σαχαραουοί να αποκτήσουν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης, δικαίωμα που έχει δοθεί σε όλους τους λαούς της περιοχής. Ο κύριος Ρωμέβα, δύο λεπτά. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εκπροσωπούς του Μετώπου Πολυσάριο γιατί είναι πραγματικά επίτευγμα η παρουσία τους εδώ και θα ήταν λάθος, σοβαρό, αν δεν τους προσκαλούσαμε. Θα ήθελα να αναφερθώ και στις χειρονομίες που έκανε τα τελευταία χρόνια το μέτωπο Πολυσάρι υπέρ της σύναψης μιας συμφωνίας για την ε, επίλυση της σύγκρουσης στη Δυτική Σαχάρα. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε αυτέ τι χειρονομίε, γιατί όταν μιλούμε για τι ευθύνε των συμβαλωμένων μερών, των εμπλεκομένων μερών, ορισμένα μέρη ανέλαβαν αυτέ τι ε, ε, υποχρεώσεις με μεγαλύτερη δέσμευση, με μεγαλύτερη πυγμή και μεγαλύτερη θυσία και υποχωρήσεις. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι, ήταν πραγματικά ε, εκνευριστική η εκστρατεία παραπληροφόρηση που είχε προηγηθεί για να αλλοιώσει το περιεχόμενο του ψηφίσματος και ήταν κατάπτυσος ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι προσπάθησαν να εμείνουν σε κομματικά συμφέροντα και να συμπεριλάβουν τέτοιου είδους ε, προβληματισμούς στο ψήφισμα. Δυστυχώς θα φύγω σε λίγο γιατί συζητούμε σε άλλη επιτροπή την απελευθέρωση ε, της ε, συμφωνίας ό,τι αφορά την διάθεση γεωργικών και ελευτικών προϊόντων από το Μαρόκο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι το Μαρόκο μπορεί να χρησιμοποιεί με τέτοιους όρους ε, τον πλούτο της ε, Δυτικής Σαχάρας όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Εγώ διαφωνώ με αυτή τη στάση του Μαρόκου και άλλοι είναι της γνώμης αυτής, γι' αυτό και πιστεύω θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι σχετικές συμφωνίες που έχουμε με το Μαρόκο. Λοιπόν, κλείνει εδώ ε, τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων ο κύριος Μέγερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό της ε, ε, Αραβικής Αχαραουιτικής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο του μετόπου Πολυσάριο. Είχαμε επεισόδια και στην ε, πόλη Ασμάρα που βρίσκεται υποκατοχή από τις στρατιωτικές μαροκινές δυνάμεις. Φαίνεται ότι με τη βία εισέβαλαν σε ένα, σε ένα Ινστιτούτο, σε μια σχολή και μάλιστα συνέλαβαν νέους Σαχαραουίτες. Έχετε πληροφορίες σχετικά. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη της κοινοβουλευτικής μου ομάδας και θα ήθελα να διαμηνήσετε στο Σαχαραουίτικο λαό αυτή την αλληλεγγύη, γιατί ο λαός σας είναι ένας λαός που αντιστέκεται με ειρηνικό τρόπο. Και θα ήθελα να τους συγχαρούμε για αυτή την ε, ειρηνική αντίσταση απέναντι σε μια δύναμη κατοχής που είναι παράνομη, που δεν έχει καμία κυριαρχία στα κατεχόμενα της Δυτικής Σαχάρας και παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν κάτι που είναι απλούστατο, δηλαδή να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο, δεν καταφέραμε να το εφαρμόσουμε χρόνια ολόκληρα τώρα στη Δυτική Σαχάρα. Και δεύτερον, ποια είναι η γνώμη σας σε ό,τι αφορά την ε, αδιαφορία της Ισπανικής κυβέρνησης ε, σε ό,τι αφορά την ε, επίσπευση της διαδικασίας αποικιοποίησης. Όλοι γνωρίζουν ότι οι συμφωνίες της Μαδρίτης ήταν παράνομες, το λένε και τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν μπορεί να διαβεβαστεί αυτή η διοίκηση σε κανένα άλλο κράτος. Αυτό λέει το δίκαιο. Και ποιος είναι ε, ποια είναι η εκτίμησή σας για το ρόλο της Ισπανίας αυτή τη σύγκρουση ό,τι αφορά την ε, εγκατάλειψη αυτής της διοίκησης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην περίπτωση αυτή και ελπίζω η Λέιδη Άστον ε, να συμπεριλάβει και το θέμα της Δυτικής Σαχάρας στο πρόγραμμα εργασιών για το προηγμένο καθεστώς που θα θέλει να δώσει το Μαρόκο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ούτσαλέκ, παρακαλώ να παραμείνετε σε ένα πεντάλεπτο στην ομιλία σας, όχι περισσότερο. Θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάντως για την ευγένειά σας. Θα έλεγα καταρχήν ως προς το πολιτικό υπόβαθρο και το πολιτικό πλαίσιο ότι Έχουμε να κάνουμε εδώ με μια δικία γιατί οι Σαχαραουίτες θέλουν να ψηφίσουν, να ψηφίσουν με δημοκρατικό τρόπο. Και πραγματικά τη σήμερα ημέρα μας συγκλονίζει να βλέπουμε πρωτεύουσες να μην ενδιαφέρονται ή να δείχνουν μια συνενοχή μεταξύ τους ε, εις βάρος της Δυτικής Σαχάρας. Η Δυτική Σαχάρα είναι πολύ κοντά στις Κανάριες νήσους. Η Δυτική Σαχάρα είναι μια όμορφη σχεδόν περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε 14.000 ε, μίλια μας χωρίζουν από, την, από το Ταγκέρι από, τη, από το Βόρειο Μαρόκο και από το Γιβραλτάρ. Το Μαρόκο έχει συνάψει συμφωνία με το μέτωπο Πολυσάριο. Και το μέτωπο Πολυσάριο έκανε πολλές υποχωρήσεις για να συναυθεί η συμφωνία αυτή το 1991. Υπάρχει αποστολή το ΙΕ στη Δυτική Σαχάρα για τη διοργάνωση του δημοψηφίσματος. Αλλά το δημοψήφισμα δεν γίνεται επειδή δεν θέλει το Μαρόκο. Ο Χασάν ο δεύτερος, ο πρώην βασιλέας του Μαρόκου, μέχρι το 1999 ποτέ δεν είπε ότι είναι κατά του δημοψηφίσματος. Απλώς ε, δημιούργησε εμπόδια στη διεξαγωγή του. Και μάλιστα έκανε ό,τι μπορούσε για να το κερδίσει κιόλα, γιατί μετέφερε πολλούς Μαροκινούς, χιλιάδες Μαροκινούς από το Μαρόκο, τους μετεκατέστησε στα κατεχόμενα εδάφη για να εξασφαλίσει υποστήριξη στο δημοψήφισμα. Η τωρινή κυβέρνηση όμως είπε ρητά ότι όσο έχουμε συμφωνία δεν θα γίνει δημοψήφισμα. Αυτή είναι μια κατάφορη αντίφαση, κύριε Πρόεδρε, μεταξύ του τι συμβαίνει στη Δυτική Σαχάρα και του τι συμβαίνει στο Νότιο Σουδάν, για παράδειγμα, σήμερα. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θέλουν οι συμφωνίες μεταξύ της Σουδανικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης του Νότου να εφαρμοστούν αμέσως. Ενώ στη Δυτική Σαχάρα έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια που το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει ε, πει ότι από τη στιγμή που το Μαρόκο δεν θέλει ψήφισμα, ε, δημοψήφισμα να μην γίνει δημοψήφισμα, επειδή υπάρχουν διαφωνίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι Σαχαραουίτε δεν είναι κατά του Μαρόκου. Είμαστε μια μικρή χώρα που θέλει να ζήσει ειρηνικά και θα θέλαμε να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα στη ζώνη αυτή. Είμαστε η μοναδική χώρα της ζώνης του Μαγκρέπ που δεν αναγνωρίζει τα σύνορα των γειτόνων του Μαρόκου. Δεν αναγνωρίζονται τα σύνορα ούτε με το Μαρόκο, ούτε με την Αλγερία, ούτε με την Ισπανία. Και για πάνω από 15 χρόνια διεκδικούνται και η Μαυριτανία και ένα τμήμα του Μαλή από το Μαρόκο. Αν το Μαρόκο δεν αναγνωρίσει τα σύνορα, αν δεν αναγνωρίζει τα σύνορα των γειτονικών της χωρών, δεν πρόκειται να, να αποκατασταθεί η ειρήνη. Τώρα τι προοπτική υπάρχει για την σύσταση Διεθνούς Ερευνητικής Επιτροπής για να διαλευκανθεί η κατάσταση. Γιατί το Μαρόκο απελάβει τους πάντας αυτή τη στιγμή. Και για να απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνατε, πόσα θύματα έχουμε και τι στοιχεία υπάρχουν ή τι έγινε με αυτή τη δολοφονία στο, στο Λαγιούν. Εκ μέρους του μετόπου Πολυσάρη δεν μπορώ να σας δώσω ακριβή στοιχεία για το τι συνέβη. Ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Φανταστείτε, ένας καταβλισμός άμαχο πληθυσμού με 25-30 χιλιάδες ανθρώπους στις 6 τα χαράματα βρίσκεται αντιμέτωπος απέναντι σε δεκάδες χιλιάδες στρατιωτών που ήρθαν από το Μαρόκο και απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις, στις δυνάμεις ασφαλείας ο πληθυσμός αυτός προσπάθησε να ξεφύγει προς το Λαγιούν και είχαμε τετραήμερη καταστολή. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσοι γύρισαν στα σπίτια τους και πόσοι αγνοούνται. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι ζωντανοί ή πόσοι είναι νεκροί. Κανείς δεν μπορεί να δώσει τέτοια στοιχεία, ούτε καν οι δημοσιογράφοι που το τελευταίο τρίμερο ε, έμεναν στο Λαγιούν. Και αυτοί εκδιώχθηκαν, πελάθηκαν χθες. Κανείς δεν μπορεί να δώσει με ακρίβεια τα στοιχεία. Γιατί το Μαρόκο δεν θέλει. Σκοτώνει καθημερινά τους Σαχαραουίτες. Έχουμε κατάσταση πολιερκίας αυτή τη στιγμή στο Λαγιούν. Σε ό,τι αφορά το νομικό καθεστώς. Τα... Ο ΙΕ θεωρεί την Ισπανία ως ε, διοικούσα δύναμη. Μόνη της Ισπανία δεν μπορεί να λέει νίτο τα μου εγώ αποχώρησα το 76 και δεν φέρω καμία ευθύνη. Έχει ευθύνη η Ισπανία απέναντι στον ΟΗΕ και πολιτική και ηθική ευθύνη να διεκπαιρεώσει τη διαδικασία αυτοδιάθεσης του σαχαραουίτικου λαού και διεξαγωγής δημοψηφίσματος. Δεν μπορεί να απεκδίεται των ευθυνών της η Ισπανία. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Χθε, μάλιστα, η έπικη και η ε, στρατιωτικές μαροκινές δυνάμεις εισέβαλαν σε σχολεία στη Σμάρα και στη Λαγιούν χτυπώντας τον κόσμο και καταστρέφοντας τα πάντα. Γίνεται μια απόπειρα εθνοκάθαρσης αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια απόλυτη ρήξη μεταξύ των Σαχαροϊτών των κατεχόμενων και του Μαρόκου. Θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πιο δραστήριο ρόλο στην περιοχή. Θέλουμε να διορίσετε ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Σαχάρα, στη ζώνη, για να συμβάλλει άμεσα στη διεθέτηση της σύγκρουσης. Θέλουμε ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα προς το Μαρόκο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι και προς το συμφέρον του Μαρόκου να, διεκπερα... να περατωθεί αυτή η σύγκρουση να τεθεί ένα τέλος, ένα δημοκρατικό τέλος σε αυτή τη διένεξη για να μπορέσει και ο σαχαροίτικος λαός να ασκήσει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ δυστυχώς να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να μειώσω περαιτέρω σε ένα λεπτό τις ομιλίες των επομένων ομιλών. Κύριος Μιγιάν ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους του με το Πολυσάριο που ήρθαν για να μας δώσουν τη δική τους εκδοχή των επεισοδίων. Γιατί δεν διαλύθηκε ειρηνικά ο καταβλισμός, για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε η βία, γιατί ε, οι Μαροκινοί δίνουν άλλη εκδοχή, ότι υπήρχαν ε, εγκληματίες στον καταβλισμό. Ποια είναι η δική σας ε, παραλλαγή. Γιατί μας είπατε και για αγνοούμενους, για δολοφονίες, για νεκρούς και μία ερώτηση για το μέλλον. Ποιο είναι το μέλλον των άτυπων συνομιλιών που γίνονται στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ σε μια τόσο τεταμένη και έκριθμη κατάσταση. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό βαρνιό. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την οργάνωση αυτής της ακρόασης Λυπάμαι που ο Υπουργός Εξωτερικών του Βασιλείου του Μαρόκου δεν δέχθηκε την αρχική σας πρόταση. Γιατί νομίζω ότι το να υπάρξει διάλογος ανάμεσα στην Αλγερία και το μέτωπο θα ήταν ένα βασικό θα έλεγα στοιχείο που θα ευνοούσε να βρεθεί κάποια λύση σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στη Σαχάρα. Είχα πάει στο Λαγιούν ε, πρόσφατα δεν είδα αυτά τα οποία άκουσα από πλευράς του μετόπου Πολυσάριο τώρα. Δεν μπόρεσα να πάω όμως στο Τιντούφ και θα ήθελα να μου πείτε γιατί δεν υπάρχει σήμερα από πλευράς της ΥΠΑ της Αρμοστίας η δυνατότητα καταγραφής με διαφανή τρόπο των κατοίκων των καταβλισμών του Τιντούφ. Είναι απαραίτητο η απογραφή αυτή να ολοκληρωθεί. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις στο γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να συνεχιστεί το πρόγραμμα οικογενειακών επισκέψεων, ένα αυστηρά ανθρωπιστικό πρόγραμμα. Άκουσα χτες ότι ο Μουστάφα Σαλμά απελάθηκε στη Μαυριτανία από το Πολυσάριο. Εκπλήσωμε για την απέλαση αυτή, η οποία και νομικά και ανθρωπιστικά δεν ανταποκρίνεται στη Σύμβαση της Γενέβης του 1951. Να διευκρινίσω κύριε Παρνιό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλγερίας απάντησε χτες λέγοντας ότι δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί έχει άλλες υποχρεώσεις αλλά απάντηση δόθηκε, δεν είναι ότι δεν δόθηκε καμία απάντηση. Κυρία σε ένα λεπτό. Νομίζω ότι η βαναυσότητα της επίθεσης αυτής εκ μέρους του Μαρόκο είναι συγκλονιστική. Και μάλιστα προσπαθήσαμε να πάμε εκεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει να στείλουμε νέα αποστολή στο Λαγιούν για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για το τι συνέβη πραγματικά θα πρέπει το Μαρόκο να λογοδοτήσει για τους νεκρούς, τους τραυματίες και τους αγνοούμενους. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε απέναντι σε αυτή την σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα. Γιατί είναι ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι θέμα του δικαιώματο αυτοδιάθεση του σαχαροϊτικού λαού. Πρόκειται για μια γειτονική περιοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι προ το συμφέρον μα να επιληθεί αυτό το θέμα. Και δεν μιλώ για τον πλούτο τη Δυτική Σαχάρα που δεν τις εκμεταλλεύεται ε, ο σαχαραοίτικος λαός. Είναι προς το συμφέρον όλων των ε, χωρών της περιοχής, γιατί ε, δεν έχουμε μόνο την Ελία, έχουμε και το πετρέλαιο, έχουμε φυσικούς πόρους. Και επίσης έχουμε και μια ζώνη στην οποία δρούν και εγκληματίες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κλείουμε τα μάτια απέναντι στη Δυτική Σαχάρα. Και έχουμε το καλό παράδειγμα του Ανατολικού Τιμόρ, που είναι πλέον παράδειγμα προς για καλή γειτνίαση με την Ινδονησία. Παρόλο που και αυτή η χώρα ε, για ένα διάστημα είχε παράνομα και στρατιωτικά εισβάλλει στην περιοχή. Παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο σας γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει και πρέπει να απαντήσει ο κ. Ολτσάλεκ. Μπέναρα του. χαιρετίζω την παρουσία σας. Πράγματι η κατάσταση στην Σαχάρα είναι περίπλοκη και δεν μπορεί κανείς να έχει μια ξεκάθαρη θέση. Είναι δραματικό το ότι ίσως ε, μια δεκάδα ε, ε, κατοίκων της περιοχής έχασε τη ζωή της και δεν ήταν προφανώς μόνο Μαροκινή. σχετικά με τις δυνατότητες που θα έδιναν την ελευθερία, την αυτοδιάθεση στον λαό των Σαχαραουή. Υπάρχει άλλος τρόπος από το δημοψήφισμα, εφόσον το δημοψήφισμα δεν είναι εφικτό. Είπατε ότι είσαστε για ένα ε, ευημερών και ε, ε, ευτυχισμένο Μαγκρέμπ. Τι θα κάνετε εφόσον όμως το δημοψήφισμα δεν είναι εφικτό. Τελευταίος ομιλητής Παντσέρη, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για το Μαγκρέμπ. Έχει σημασία η παρουσία σήμερα του εκπροσώπου του μετόπου Πολυσάριο. Το ψήφισμα που έχουμε μπροστά μας είναι ένα ψήφισμα το οποίο δείχνει τη συγκλίνουσα αντίληψη που χαρακτηρίζει τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ψήφισμα αυτό καταδικάζει τα γεγονότα, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα, και απευθύνει έκκληση σε όλους να προχωρήσουν σε κάποια βήματα με πρωταγωνιστή φυσικά τον ΟΗΕ. Δεν μας διαφεύγουν οι συσχετισμοί δυνάμεων στην περιοχή, τα προβλήματα των ε, Σαχαραουή, όπως επίσης και η λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων της περιοχής. Θα θέλαμε την άποψή σας λοιπόν για όλα αυτά ε, εφόσον μπορούμε να διασφαλίσουμε κάποιες προϋποθέσεις για να πετύχουν οι διαπραγματεύσεις. Καταρχάς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε περιφερειακή βάση το πρόβλημα και το θέμα της Αλγερίας δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεύτερο στοιχείο είναι το να σταματήσουν όλες οι μονομερείς ενέργειες και ε, προκλήσεις από όλες τις πλευρές. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί σύντομα εφόσον θέλουμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Τέλος, ίσως να υπάρξει, κύριε Πρόεδρε, μία αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία να μπορέσει να έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα ε, επιτόπου μια αντιπροσωπεία χωρίς προκαταλήψεις η οποία να ελέγξει το τι συμβαίνει εκεί έτσι μόνο η λύση θα βρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνίστρια. Ευχαριστώ κύριε Παντζέρη. Παρακαλώ πέντε λεπτά όχι περισσότερο κύριε Ολτσαλέκ γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο. Με ρώτησε κάπως, κάποιος γιατί καταστράφηκε ο καταβλισμός. Μα, εκεί είναι το πρόβλημα μια ειρηνική διαδήλωση, μια ειρηνική διαμαρτυρία που κράτησε ένα μήνα και, και μάλιστα οι οργανωτές ε, είχαν ε, χρονοβόρες διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για ένα ολόκληρο μήνα και τώρα το Μαρόκο τους κατηγορεί, κατηγορεί τους διοργανωτές αυτής της διαδήλωσης ως συμμορία εγκληματιών. Και μάλιστα θα τους πάει και στρατοδικείο. Μετά από ένα ολόκληρο μήνα διαπραγματεύσεων που είχε μαζί τους. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος της μαροκινής κυβέρνησης πολλές φορές έκανε δηλώσεις στην τηλεόραση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δηλώνοντας ότι έχουμε διαπραγματεύσεις με τους αδελφούς μας που έχουν κοινωνικές ε, ε, δίκες, κοινωνικές ε, διεκδικήσεις και παραδεκτές διεκδικήσεις και από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει στάση το Μαρόκο. Έτσι έχει κατάσταση. Διαπραγματεύσεις. Δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα με το Μαρόκο. Γιατί το Μαρόκο δεν θέλει διαπραγμάτευση. Το Μαρόκο δεν θέλει διαπραγμάτευση. Θέλει να επιβάλλει τη θέση του. Η πρόταση για την αυτονομία έγινε δεκτή ως ε, εναλλακτική λύση από το 2003 από το μέτωπο Πολυσάριο. Όταν ο Μπέικερ είχε υποβάλει την πρότασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Τότε το μέτωπο Πολυσάριο είχε πει ναι. Δεν έχουμε καμία, κανένα πρόβλημα με την πιθανότητα της αυτονομίας. Αλλά όχι να μας επιβάλλει τη θέση του το Μαρόκο αποκλείοντας τις υπόλοιπες εναλλακτικέ λύσεις. Όπως είπα, στα νότια του Σουδάν, στο δημοψήφισμα του Νοτιού Σουδάν, θα ψηφίσουν μόνο αν θέλουν να γίνουν τμήμα του Σουδάν. Δεν έχει νόημα αυτό. Το δημοψήφισμα που δέχτηκε το 1991 το Μαρόκο μετά από 17 ετή πόλεμο είναι ένα δημοψήφισμα που θα επιτρέπει στο σαχαρίτικο λαό να επιλέξει αν θέλει την ανεξαρτησία ότι προτιμά να είναι τμήμα του Μαρόκου. Δεν θέλει όμως διαπραγμάτευση πια το Μαρόκο, θέλει απλώς να μας επιβάλλει τη θέση του. Εμείς συμμετέχουμε για να βοηθήσουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Συμμετέχουμε στο διάλογο, ένα διάλογο όμως που δεν θα πάει μακριά, αν συνεχίσουν ορισμένοι να υποστηρίζουν πάση τη θυσία το Μαρόκο. Στα γαλλικά τώρα. Έχω σπουδάσει στη Γαλλία και θα συνεχίσω στα γαλλικά. Σέβομαι τη Γαλλία, σέβομαι τα γαλλικά πανεπιστήμια και τον γαλλικό λαό με την τεράστια ιστορία. Πράγματι ο Αλγερινός Υπουργός δεν είναι εδώ σήμερα. Αν του ζητούσατε να έλθει θα πρέπει να ζητήσουμε και από την κυρία Μαριλιώτ, γιατί η Γαλλία υποστηρίζει το Μαρόκο και το εξοπλίζει. Και το λέω αυτό με κάθε διάθεση ειλικρίνειας. Η Αλγερία υποστήριξε το μέτωπο Πολυσάριο, το υποστηρίζει πάντα, δεν το κρύβει. Το ίδιο έκανε και με τη Σουάπο στην Αμιμπία και με το κίνημα στο Τιμόρ υποστήριξε και υποστηρίζει πάντα τους Παλαιστινίους, πάντα το κάνει αυτό και έχει σύνορα με το Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα. Είναι σαν η Γαλλία να μην δέχεται μια γειτονική της χώρα, η οποία κατέχει μια άλλη χώρα. Λοιπόν, είναι στη στρατηγικό συμφέρον της Αλγερίας, πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μην δέχεται το status quo που θέλει να επιβάλλει το Μαρόκο. Γιατί δεν έκανε την απογραφή η ύπατη αρμοστία, αγαπητέ φίλε, το έκανε αυτό. Οι οικογενειακές επισκέψεις στο Μαρόκο θέλει να διακρίνει ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να το κάνει και μπλοκάρει. Παρότι υπάρχει ε, συμφωνία ανάμεσα στο Πολυσάριο και το Βασίλειο του Μαρόκου για τις οικογενειακές επισκέψεις. Το θέμα του αστυνομικού που δεν είναι ο αρχηγός της αστυνομίας, είναι ένας απλός αστυνομικός, ο Σέλμα. Ο Σέλμα πήγε στο Μαρόκο, έφυγε, δικαίωμά του, αλλά οι μαροκινές υπηρεσίες οργάνωσαν ένα σοου γύρω από την περίπτωσή του. Το μέτωπο ο Πολυσάριο τον φυλάκισε πράγματι όχι γιατί είχε δηλώσει ότι είναι κατά της αυτονομίας, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με την αυτονομία, αλλά γιατί είναι αστυνομικός. Ένας Γάλλος αστυνομικός, ο οποίος θα πάει σε μια χώρα εχθρική της Γαλλίας και χρησιμοποιηθεί από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτής, της βάρος της χώρας του, προφανώς ε, υφίσταται κυρώσεις και γι' αυτό συνελήφθη από την πρώτη μέρα είναι σε επαφή με την ύπατη αρμοστία και είναι αυτός ο οποίος δέχτηκε να πάει στη Μαύρη Ιτανία. Η οικογένειά του δεν θέλει να φύγει μαζί του. Ελάτε ε, να συζητήσετε με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του αν θέλουν να φύγουν μαζί σας για να πάνε στον Σαλέ, ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Επίσης δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είστε καλοδεχούμενοι στις απελευθερεμένες περιοχές και στα στρατόπεδα καταβλισμούς προσφύγων. Αλλά θα θέλαμε ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, πράγματι να συστήσει μια αντιπροσωπεία και να έρθει και στο Αγίον σήμερα Ελάτε εσείς να δείτε πώς είναι η κατάσταση, να πάτε στις οικογένειες, στο Αλαγιούν και στη Σμάρα. Για την υπόθεση της Σμάρα που κάποιοι από αυτούς, ε, ε, κάποιοι από σας αναφέρθησαν, θα ήθελα να πω στην κυρία Γκομές ότι συγχαίρουμε την Πορτογαλία γιατί η Πορτογαλία και το λέω αυτό ανέλαβε τις ευθύνες που είχε σε σχέση με το Τιμόρ και θα θέλαμε και η Ισπανία και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών να πει ξεκάθαρα ότι πρέπει να οργανωθεί το ταχύτερο δυνατόν το δημοψήφισμα. Είναι η μοναδική λύση. Μια άλλη κυρία μου έθεσε το ερώτημα γιατί αν δεν μπορεί να οργανωθεί το δημοψήφισμα, γιατί να μην οργανωθεί το δημοψήφισμα, να σας πω κάτι λίγο αστείο. Το ανέκδοτο προτείνει την αυτονομία, λέει θα το θέσουμε σε ψηφοφορία. Από τη μία λέει ότι δεν μπορούμε να οργανώσουμε το δημοψήφισμα, ενώ κάνει μια δική του πρόταση την οποία λέει ότι θα βάλει σε δημοψήφισμα. Αυτό είναι αντίφαση. Και γιατί ο λαός των Σαχαραουί να είναι ο μοναδικός λαός των κόσμο στον οποίο αρνούμεθα την δυνατότητα να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του και να ψηφίσει. Γιατί αυτό. Λένε ότι πολλαπλασιάζονται οι μικρές χώρες. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μέλος της Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας, αναγνωριζόμαστε από 80 χώρες του κόσμου και είμαστε γεωγραφικά και δημογραφικά μεγαλύτεροι από 30 χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών και στον αραβικό κόσμο και στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό και σε άλλες περιοχές, ακόμα και στην Ευρώπη. Δεν είναι δικαιολογία λοιπόν αυτή. Δεν βλέπουμε γιατί για άλλους δεν πειράζει να είναι μικρή χώρα, ενώ για κάποιους άλλους είναι πολύ κακό. Λοιπόν, για τους Μαροκινούς και το δημοψήφισμα. Καλά. Ε, μου λέτε να σταματήσω, σταματώ. Λυπάμαι αλλά δεν υπήρξε περισσότερος χρόνος για να ακούσουμε και τα άλλα θέματα και άλλες απαντήσεις. Ξέρετε ότι η σημερινή συνάντηση αποφασίστηκε μαζί σας και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου σε μια φάση όπου είχαμε και άλλες υποχρεώσεις και γι' αυτό μας υποχρεώνει η κατάσταση να μην έχουμε πιο πολύ χρόνο. Εν πάση περιπτώσει θα συνεχιστούν οι προσπάθειες, ελπίζω να συλλέξατε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις από τους συναδέλφους. Σας ευχόμαστε κάθε τι καλό για το μέλλον και το ίδιο θα κάνουμε και με τον ομόλογό σας που θα ακολουθήσει. Grazie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 Λοδωρό. Bene, eh, ευχαριστώ, ευχαριστώ γιατί φεύγετε γρήγορα και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση. Είπα και πριν ότι ο χρόνος μας είναι πολύ μετρημένος. Έχουμε στην Επιτροπή μας και εκπροσώπους της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ιράκ και παρακαλώ τον κύριο Στίβενσον να καθίσει μαζί μας στο Προεδρείο. Όπως ξέρετε έχουμε την χαρά να υποδεχθούμε στην Επιτροπή μας τον ειδικό εντεταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ, τον κύριο Αρτ Μέλκερτ. Η παρουσία του πραγματικά είναι πολύ επίκαιρη, δεδομένων των εξελίξεων που έλαβαν χώρα το τελευταίο καιρό στο Ιράκ. Πριν από δύο εβδομάδες η Ιρακινή Βουλή ε, επανεπιβεβαίωσε τον Τζαλάλ Ταμπάνη στη θέση του Πρόεδρου Δημοκρατίας και πριν από τέσσερις μέρες ο Πρόεδρος Ταλαμπάνη ανέθεσε στον Πρωθυπουργό Αλμαλίκη να συνεχίσει τις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης. Ο Σάμα Νουιεγέφη του συνασπισμού Αράλ Αλνταγιάουι ανακηρύσσεται πρόεδρος του, Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Ιρακινού συγγνώμη, Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο του Ιράκ αυτή τη στιγμή. Κάτι που δημιουργεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία μετά από ένα εννιάμενο πολιτικού αποκλεισμού μετά τη δεξαγωγή των εκλογών. Ευελπιστούμε ότι με τη συμφωνία αυτή θα ενισχύσουμε τη σταθερότητα των ε, Ιρακινών θεσμών προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και ευημερία σε αυτή τη μαρτυρική πραγματικά χώρα. Η σταθεροποίηση του Ιράκ ε, ήταν ανέκαθεν προτεραιότητα σύσσωμης της παγκόσμιας κοινότητας και η απόσυρση των Αμερικανικών ε, στρατητικών δυνάμεων από το Ιράκ που έχει προβλεφθεί για το επόμενο καλοκαίρι Ελπίζουμε ότι δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, ανυπέρβλητα προβλήματα στις ε, Ιρακινές θεσμικές ε, δυνάμεις που θα αντιμετωπίσουν πολύ άριθμα προβλήματα ασφάλειας, ε, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στις προσπάθειες ανασυγκρότησης του Ιράκ και Υπάρχουν πολλά κοινοτικά προγράμματα εκεί. Το 2003 μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε με πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια αναπτυξιακή και ανασυγκρότησης. Μάλιστα η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί επιβεβαιώθηκε με μια συμφωνία εταιρική σχέσης και συνεργασίας με την Ιρακινή κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκε την επίσημη αίτηση για τη διαδικασία σύμφωνης γνώμη, και μάλιστα ο κύριος Μάουρο θα είναι ο εισηγητή για το θέμα αυτό. Πριν δώσω το λόγο στον ειδικό εντεταλμένο του Γενικού Γραμματέα στο ΙΕ, τον οποίο θα ακούσουμε με ιδιαίτερη προσοχή, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής ε, στο προσωπικό της Σουνάμι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματικά συνέβαλαν τα μάλα σε αυτές τις δύο δύσκολες στιγμές ε, για να εξασφαλιστεί η ευημερία του Ιρακινού λαού. Παρακαλώ κύριε Ατμέλκερ, έχετε το λόγο αν μπορείτε να περιοριστείτε σε ένα δεκάλεπτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και εξώματος των συναδέλφων που εξακολουθούν να εργάζονται κάτω από δύσκολες ακόμα συνθήκες στο Ιράκ σε καταστάσεις στις οποίες υπάρχει μια σταδιακή πρόοδος αλλά υπάρχουν και οι υπαναχωρήσεις της κατάστασης συνεχώς. Παρ' όλα αυτά το Ιράκ έχει φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό στάδιο της εξέλιξής του και είναι πραγματικά τιμή μου που μπορώ σήμερα να σας παρουσιάσω κάποιες ιδέες και κάποια γεγονότα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα κράτη-μέλη εξακολουθούν να παραμένουν στενά δεσμευμένα για την πανικοδόμηση του Ιράκ και για την πρόθεση της ολοκλήρωσης στην περιοχή και γενικά μεταξύ της Ευρώπης και αυτού του τόσο σημαντικού τμήματος του κόσμου. Θα ήθελα να κάνω ορισμένε παρατηρήσει όσον αφορά την πολιτική διαδικασία που ήταν η πιο σημαντική στο έτος που ολοκληρώνεται τώρα, αρχίζοντας πριν από ένα χρόνο με την οθέτηση του εκλογικού νόμου, μετά από μια μακρά και δύσκολη διαδικασία, να υπάρξει τελικά συνένεση πάνω στον ε, ε ελεκτικό αυτό νόμο, πρώτη φορά, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για πρώτη φορά μπόρεσε έτσι να οργανωθεί μια ομαλή μετάβαση από μία εκλεγμένη κυβέρνηση σε μία άλλη και εν αντιθέσει από ό,τι είχε γίνει την περασμένη φορά χωρίς άμεση εμπλοκή της Αμερικανικής ιδίω πλευράς. Αυτή ήταν η σημασία της οθέτησης του εκλογικού νόμου. Κατόπιν είδαμε μία εκλογική εκστρατεία, η προεκλογική εκστρατεία αν θέλετε πολύ πιο ανοιχτή από ό,τι ποτέ στο παρελθόν. Σημειώθηκαν διάφορα συμβάντα βέβαια, τα οποία όμως δεν είχαν επιπτώσεις στην συμμετοχή στις εκλογές που της τάξης του 62-63% πολύ υψηλή πολλοί Ιρακινοί γιόρτασαν την ευκαιρία να μπορούν να ψηφίσουν. Κατά μέτρηση των ψήφων μετά χρειάστηκε αρκετό καιρό. Βασίστηκε όμως σε μια καλή διαδικασία με αξιόπιστο αποτέλεσμα. Παρόλο που υπήρχε προσφυγή κατά το αποτελέσματο και χρειάστηκε να γίνει εκ νέου καταμετρηστή και γι' αυτό τα τελικά αποτελέσματα υπήρχαν μόλις τον Μάη. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια μακρά διαδικασία δημιουργίας κυβέρνησης χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του Ιράκ. Μια ανεξάρτητη διαδικασία οργανωμένη από τα, τις χίλιες πολιτικές ομάδες όπως είναι οργανωμένη στο Κοινοβούλιο. Η διαδικασία αυτή αυτή τη στιγμή δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. Είμαι προσεκτικός πώς θα το διατυπώσω αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η διαδικασία και αναμένεται ότι ο Πρωθυπουργός Μαλική από τον οποίο ζητήθηκε από τον ε, Πρόεδρο να δημιουργήσει την κυβέρνηση θα εξακολουθεί να ηγείται της χώρας. Καταρχήν, ε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά θέματα για τα οποία συνειδητήθηκαν όλα τα σημαντικά κόμματα από τις αρχές Νοεμβρίου και μετά γύρω από τις τράπεζες και τέλος η επιλογή των υποψηφίων για τις θέσεις των υπουργών θα πρέπει επίσης να προχωρήσει. Ορισμένοι ρωτιούνται γιατί χρειάζεται τόσο καιρό. Και οπωσδήποτε για την εξέλιξη στο εσωτερικό του Ιράκ παρεμπόδισε η διαδικασία αυτή για τη συνέχιση πολύ σημαντικών ε, προσπαθειών για την επανοικοδόμηση της χώρας, οικονομικής ανάπτυξης, καταπολέμησης της στόχας, Πολλές από τις προτεραιότητες δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν στις αρχές του έτους. Από την άλλη μεριά όμως, είναι σωστό ότι δεν υπήρχε κανένα προηγούμενο για την ε, μεταβατική διαδικασία της κυβέρνησης που είδαμε να εμφανίζεται και βάσει αυτών νομίζω το κύριο επίτευγμα είναι ότι όλα τα κόμματα παρέμειναν προσκολλημένοι στην συνταγματική διαδικασία ούτως ώστε να υπάρξει η σωστή κυβέρνηση τελικά. Είναι θέμα και εικασίας Ποιε είναι οι διαφορέ μεταξύ τη νέα κυβέρνηση και της παλιάς. Ιδίω μια που φαίνεται ότι υπάρχει ε, αρκετή συνοχή στις θέσει που κατελήφθησαν ή θα καταληφθούν. Πιστεύω όμω ότι θα μπορούσε κανένας να περιμένει διαφορετική διαδικασία της εξεσρώπησης των δυνάμεων. Ότι η Σούνη θα ήταν πιο και οι σαντρίστες έχουν δυναμώσει τη θέση τους σχετικά με το παρελθόν. Εγώ νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα παίξει πιο φυσικό ρόλο στις σχέσεις του με την κυβέρνηση και τέλος δεν έχουν βέβαια ακόμα οριστεί όλε οι λεπτομέρειε, αλλά το λεγόμενο Εθνικό Συμβούλιο για την ψηλότερη πολιτική, όπω λέμε, σημαντικότερη πολιτική, θα παίξει το ρόλο του στην εξισορρόπηση για να υπάρξει μια καλύτερη ισορροπία από εκείνη που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό βέβαια δεν ξέρουμε. Είναι προσδοκία, είναι εικασία. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να περιμένουμε πραγματικά το αποτέλεσμα. Η συμφωνία για μια νέα κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν συνεχιζόμενες ανησυχίες για την κατάσταση ασφάλειας της χώρας. Η ασφάλεια βέβαια βελτιώθηκε από τα σκοτεινά έτη του 2006-2007 και εν του 2008. Παρ' αυτά, τα διάφορα επεισόδια και ο ρυθμός των σκοτωθέντων επί καθημερινής βάσης για τη διάρκεια του 2010 δεν έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την παρόμοια περίοδο του 2009, πράγμα που παραμένει ανησυχητικό. Παρ' αυτά, πολλοί παρατηρητές ε, τονίζουν έχει βελτιωθεί το δυναμικό των ε, δυνάμων ασφαλείας του Ιράκ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια να προετοιμαστούν για την κατάσταση κατά τη διάρκεια του 2011, όπου σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ του Ιράκ και των ΗΠΑ της Αμερικής, θα αποσυρθούν όλες οι αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του έτους. ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά την ασφάλεια, είναι η προσοχή που αποδίδεται στις μειονότητες, ιδίως στις χριστιανικές ε, μειονότητες βαθάκια στη Μινοβά. Και βλέπω ότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία τα προβλήματα των ε, ομάδων αυτών μειονοτήτων εδώ στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα το χαιρετίζουμε αυτό γιατί έτσι συμπληρώνουν δικέ μα μας να βρεθούν κάποιε λύσει για να μπορέσουν να προστατευτούν τα συμφέροντα των μειονοτήτων αυτών κατά των Θέλω να σα πω ότι έχουμε πρόσφατα αναλάβει την συνεργασία για το θέμα αυτό και προσπαθούμε θέμεθα να συνεχίσουμε για να βελτιώσουμε την ε, κατάσταση των μειονοτήτων. Λόγω των σημαντικών επιπτώσεων των όσων διαμήφθησαν από το 2003 και μετά, το Ιράκ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστιες ανάγκες οικονομική ανάπτυξη, εξ, ε, εξωτερικές επενδύσεις, εσωτερικές επενδύσεις κατά αποτελέμηση τη ένδυας που πλήττει περίπου το 25% του πληθυσμού. Δεν θα επιστρέφω σε λεπτομέρειε αυτή τη στιγμή, αλλά ελπίζουμε ότι αν βελτιωθεί η ασφάλεια και αν η πολιτική κατάσταση είναι πιο σταθερή, θα μπορέσει το, η κυβέρνηση να πετύχει αυτά που θέλει. Το 2011 δηλαδή θα είναι πιο επικοδομητικό προς την κατεύθυνση αυτή. Τελειώνοντα, επιτρέψτε να κάνω δύο ε, σχόλια όσον αφορά το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλο των Ηνωμένων Εθνών βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ιδίω στην 1770 του 2007, όπου προθέμεθα να βοηθήσουμε αιτήσει της κυβέρνησης του Ιράκ, ιδίω για την πρόθεση της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την πολιτική διαδικασία και την ανθρωπιστική εξέλιξη, την εξέλιξη δηλαδή στον ανθρωπιστικό τομέα. Για να το πτύχουμε αυτό, συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο και με την κοινωνία των πολιτών και θα ήθελα να τονίσω ότι η βάση της πολιτικής συμφωνίας ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας δρούμε μόνο κατόπιν πρόσκλησης της κυβέρνησης του Ιράκ. Στο μέλλον θα ασχοληθούμε κυρίως στην ενίσχυση των πολιτικών διαδικασιών που ελπίζουμε ότι θα οδηγήσουν σταθερότητα στις λεγόμενες αμφιλεγόμενες περιοχές που αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από την επίλυση των διαμάχες ε, Αράβων και Κούρδων. Επίσης ε, θα ε, έχουμε την προ, καταβάλει προσπάθειες για την βελτίωση των σχέσεων Ιράκ και Κουβάιτ, ιδίως όσον αφορά το λεγόμενο κεφάλαιο 7 και τις κυρώσεις που προβλέπετε εκεί, που ανάγονται στον πόλεμο του 1991 και όπου θα πρέπει να υπάρχει πρόοδος βάσει των διδαγμάτων του πρόσφατου παρελθόντος. Επίσης, ανθρώπινα δικαιώματα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα κάνουμε μια παρουσίαση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίω όσον αφορά καταπατήσεις των εν λόγω κανόνων. Ε, Εξετάζουμε στενά την κατάσταση στην ΑΣΑΦ Έχουμε συχνές και τακτικές επαφές με εκπροσώπους της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ανθρωπιστική κατάσταση εκεί. Αναφερόμενοι βέβαια σε μια αρχή βασική ή σε μια σειρά βασικών αρχών και τονίζω προς την Ιρακική κοινή κυβέρνηση ότι πρέπει να τη στηρίσουν. Τώρα, για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχεί για τη συνεργασία με την αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με πολλά κράτη-μέλη. Ελπίζουμε και αναμένουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει προσκολλημένη στην συνεργασία και ενίσχυση του Ιράκ. Γι' αυτό χαιρόμαστε και για την συμφωνία πλαίσιο. Και πιστεύουμε ότι αν εξετάσουμε τα οικονομικά συμφέροντα, την ενεργειακή πολιτική και τα σχετικά συμφέροντα και το συμφέρον για την προώθηση των αξιών και την ενίσχυση της κυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλά τοποθετημένη για είναι ισχυρό εταίρο του Ιράκ και εμεί θα συνεργαστούμε θεσμικά σα όργανα προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, Δ. Μέλκερτ. Το λόγο έχει ο κ. Στίβενσον, που είναι ο πρόεδρο τη Αντιπροσωπεία για τη σχέση με το Ιράκ. Δύο λεπτά παρακαλώ κύριε Στίβενσον. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας να υπάρχει αυτή η κοινή συνεδρίαση με τον κύριο Μέλκερ. Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή για μας και για τα μέλη της της Εκλογής στο Ιράκ να συμμετάσχουμε σε αυτή σας την ακρόαση. Ταυτόχρονα, εξ ονόμως στην μας, θα ήθελα να πω κι εγώ πόσο σας σεβόμαστε κύριε Μέρκε για το, το καταπληκτικό έργο που επιτελέστηκε κάτω από φοβερά δύσκολες συνθήκες. Ξέρετε ότι η αντιπροσωπεία μας ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2008 σαν μια μόνιμη αντιπροσωπεία ad hoc. Αλλά μετά τις εκλογές είμαστε τώρα ήμασταν τώρα μια πλήρης αντιπροσωπεία για τις εκλογές στο ΕΡΑΚ και εξετάζουμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο συνεργασίας με το Ιράκ, μεταξύ Ιράκ και Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, όπως είπε ο Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει πάνω από 1,094 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2003 μέχρι σήμερα για την επανοικοδόμηση του Ιράκ. Και το κάναμε αυτό γιατί έχουμε κάθε συμφέρον να επανέλθει η ειρήνη, η δημοκρατία, η ελευθερία εκεί. Γιατί θέλουμε επίσης ότι οι πρόσφυγες που έχουν φύγει μετά τον πόλεμο στις γειτονικέ χώρες, πάνω από ένα εκατομμύριο είναι αυτοί, να αισθάνονται ότι μπορούν να επιστρέψουν. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα με την παρεμπόδιση, παρενόχληση θα μπορούσαμε να πούμε, των γειτονικών χωρών προς το Ιράκ, ιδίως το Ιράν βέβαια. Χαίρομαι που αναφέρετε ότι το Ηνωμένα Έθνη λαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά το θέμα της προστασίας των μειονοτήτων. και χαιρόμαστε που είπε η κυβέρνηση ότι προστατεύσει όχι μόνο τις ε, μειονότητες όπως τους χριστιανούς αλλά και άλλες μειονότητες που έτυχαν πιέσεων τους τελευταίους μήνες. Κύριε Μέλκερ, γνωρίζετε σίγουρα ότι την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ενέκρινε το Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα για το, τη δανειτική ποινή και για τους φόρους στους χριστιανούς στο Ιράκ. Και θα μπορούσαμε επίσης να διακόψουμε την ε, χρήση της θανατικής ποινής στο Ιράκ. Μεγάλη πλειοψηφία των μελών, 401 για να είμαι ακριβής, υπέγραψαν μια γραπτή διαμαρτυρία. Χάρηκα που το αναφέρατε στα σχόλιά σας εισαγωγικά. Ανησυχούμε ιδιαίτερα που Άσραφ βρίσκεται σε πολιορκία, οι άρρωστοι δεν μπορούν να έχουν φάρμακα, δεν μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία. Υπάρχουν ε, δεν ξέρω πώς μεγάφωνα που συνεχώς εκπέμπουν ε, προπαγάνδα 24 ώρες το 24 ώρο Όλα αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στους ανθρώπους αυτούς. Υπήρχαν κάποιες φήμες, κύριε Πρόεδρε, στις αρχές της εβδομάδας ότι ο Ιρακινός στρατός ετοιμάζει μια επίθεση κατά του κατευρισμού του Άσραφ. Ελπίζω κύριε Μέλκερ να μπορείτε να κάνετε τα πάντα δυνατό για να αποτραπεί μια τέτοια επίθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ελπίζω το λόγο ο κύριος Μάωρο, ο εισηγητής μας για το Ιράκ. Ευχαριστώ. Και λιγότερο από δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε. Γιατί νομίζω όλα τα θέματα τέθηκαν επιτάπητος. Θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες για δύο θέματα. Ρόλος των κυβερνήσεων στην προσπάθεια αποσταθεροποίησης του Ιράκ. Ποια είναι η γνώμη του δόκτωρα Μέλκερτ. Υπάρχει στρατηγική του ΟΗΕ ως προς το θέμα αυτό. Γιατί τουλάχιστον τέσσερι σημαντικοί και μεγάλοι γείτονες του Ιράκ προσπαθούν ε, συστηματικά να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. άφησαν τη δρομοκρατία και κάνουν ένα διπρόσωπο παιχνίδι Και νομίζω ότι θα μπορούσε η παγκόσμια κοινότητα να συνειδητοποιήσει αυτό το φαινόμενο. Το θέμα των χριστιανών δεν είναι ένα κοινό ζήτημα μειονότητας. Και μάλιστα είχαμε και τη δίωξη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Και αυτό συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση του Ιράκ. Ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα, σε πολλά χριστιανικά χωριά, οργανώθηκε ένα είδος αντάρτικου. Υπάρχει λοιπόν στρατηγική του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και μάλιστα είχαμε την πρόταση του Ταλαμπάνη να συγκεντρώσει όλους τους χριστιανούς σε μία και μόνο επαρχία για να επιλύσει το πρόβλημα με τον τρόπο αυτό. Για πέντε λεπτά το λόγο έχει ο Δ. Μέλκερτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Στίβενσον και την αντιπροσωπεία του για το ε, ενδιαφέρον που δείχνουν στις εξελίξεις στο Ιράκ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Και προβλέπουμε σε μια συνεχή συνεργασία μαζί σας οπωσδήποτε σημειώνουμε τις ανησυχίες που υπάρχουν, ιδίως στο καταβλισμό ΣΡΑΦ. Αυτό που κάνουμε εμείς, Σουνάμι, είναι να ελέγχουμε την κατάσταση με εβδομαδιαίες επισκέψεις στο καταβλισμό, με συζητήσεις με όλους, ακόμα και εκπροσώπους των εκεί κατοίκων, και με την μεταβίβαση των ε, εντυπώσεων και ανησυχιών μας στην Επιτροπή Ασραφ, ε, που είναι μια διευπουργική επιτροπή στη Βαγδάτη που ασχολείται με το θέμα του Ασραφ. Επίσης, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, για να έρθουμε σε επαφή με το, τους εκπροσώπους των κατοίκων στην περίπτωση που χρειάζεται αυτό, αν υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, ενημερωνόμαστε εμείς και εμείς ενημερώνουμε εμείς τις αρχές, χωρίς βέβαια να αποκρίτουμε την ησυχία μας. Αναφερθήκαν αυτά τα μεγάφωνα, παραδείγματος χάρη. Και εγώ συμφωνώ ότι αυτοί οι, αυτά τα μεγάφωνα δεν έχουν καμία λογική ε, αποστολή και γι' αυτό έχουμε ζητήσει να αποσυρθούν. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Όπου προσπαθούμε όσο μπορούμε να παρουσιάσουμε απόψεις που βασίζονται στις βασικές αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σαν κατευθυντήριες αρχές για την κατάσταση αυτή. Αυτό είναι βέβαια η πρακτική αντιμετώπιση αν θέλετε. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η πολιτική. Η κυβέρνηση έχει εκφράσει την βούλησή της και προωθούμε εμείς συνεργασία μεταξύ της ε, κυβέρνησης του Ιράκ και κατά των περισσότερων άλλων κυβερνήσεων που εκπροσωπούνται στο Ιράκ για να δούμε πώς θα επιληθεί το θέμα που είναι οπωσδήποτε πολύ προβληματικό. Θέλουμε να στοιχήσουμε κατεύθυνση αυτή και προσβλέπουμε και τι δικέ μα απόψει. Όσον αφορά τώρα τι παρατηρήσει του κυρίου Μάουρο, θα κατανοείτε ότι ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών δύσκολα μπορεί να σχολιάσει το ρόλο κάποιων κρατών μελών. Γι' αυτό θα περιοριστώ στο να σας πω απλώς ότι είναι στα πλαίσια της εντολής μας να προωθούμε τις διασυνδέσεις μεταξύ του Ιράκ και των γειτονικών χωρών. βάσει βέβαια επικοδημητικών ε, ε, μέτρων για τα οποία έχει κάθε συμφέρον το Ιράκ. Τώρα, τι έχει παρατηρηθεί γύρω από την πολιτική διαδικασία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο συνεργασίας. Πολλοί εκπρόσωποι του Ιράκ πήγαν σε διάφορες πρωτεύουσε και υπάρχουν κάποιες δηλώσεις όσον αφορά τις προτιμήσεις ε, πολιτικών για την πολιτική διαδικασία. Όλα αυτά μπορούν απόλυτα να είναι τμήματα μιας επικοδομητικής δέσμευσης. Υψηλά επίπεδα δηλαδή συνεργασίας με τις γύρω περιοχές. Δεν υπάρχει νομίζω αμφιβολία ότι μεταξύ των επιπτώσεων των ε, ε, διασυνδέσεων αυτών και των προσπαθειών του ΟΗΕ όλοι οι γείτονες να συμμετάσχουν σε αυτή την τόσο επικοδομητική ε, ημερήσια διάταξη σε αυτά τα επικοδομητικά και ασφαλή πλαίσια καταβάλω προσπάθησε να προωθηθεί κατά το δυνατόν η οικονομική κατάσταση. Για τους χριστιανούς οι παρατηρήσεις που κάνετε ήταν σωστέ. Εμείς ερχόμαστε σε επαφή με όλους και με τον πρόεδρο Ταλαμπάνη για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εμείς προωθήσαμε την ε, ε, έγκριση ενό κανόνα δε μήνυμα για τις μειονότητες. Είμαστε σε επαφή και με τους προσώπους του Συμβουλίου όπου η ανησυχία σας βρίσκουν ανταπόκριση. Προσπαθούμε να βρούμε μια βάση οι χριστιανοί να συμμετάσχουν στην κοινωνία αυτή. Μια κοινωνία που έχει πολλή εμπειρία πώς μπορούν οι διάφορες εθνότητες να συνεργάζονται. Μόνο τα τελευταία χρόνια διακυβεύτηκε αυτό. Και αυτό είναι ανησυχητικό όχι μόνο για τους χριστιανούς, αλλά και για τους χριστιανούς. Ε, Ένα λεπτό Γκόμες. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μάλκερ και τον προκάτοχό του για την τεράστια προσπάθεια την οποία έχουν κάνει. Θα ήθελα να τον ρωτήσω να μου πει καταρχάς αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πάει στα γραφεία της και μπορεί να μετακινείται ελεύθερα σε επίπεδο ασφαλείας ενώ γιατί αυτό δεν συνέβαινε όταν επισκέφτηκα εγώ το 2008 την Βαγδάτη. Το να έχει τις δικές της εγκαταστάσεις φυσικά είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μου πείτε επίσης αν η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται αποδοτική στον τομέα της αποκατάστασης των θεσμών, του κράτους δικαίου και γενικότερα στο θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών και επίσης ε, έχετε επαφές με τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις για το εμπορικό κομμάτι. Είδαμε ότι ο Γάλλος Υπουργός Εμπορίου είχε πάει πρόσφατα εκεί. Πώς είστε. Αλλά διαρωτώ με τι ακριβώς ε, αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το διακύβευμα ιδιαίτερα στον τομέα του φυσικού αερίου. Αρλάκι ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τους ε, χριστιανούς και τους διωγμούς εις βάρος των χριστιανών. Ε, είναι οι μοναδικές διώξεις που υφίστανται θρησκευτικέ μειονότητες ή υπάρχουν ε, πολλαπλές τέτοιου είδους φιλετικές θρησκευτικές βίες ενέργειες και γιατί. Ξαφνικά αυτό το θέμα ξεκίνησε τον τελευταίο καιρό, ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχε τόσο πρόβλημα. Τώρα για την ανοικοδόμηση του Ιράκ, διεθνής βοήθεια. Δεν είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τον τρόπο με τον οποίο δίδεται η διεθνής βοήθεια στη χώρα του Αφγανιστάν. Το ίδιο ισχύει επίσης και για το Ιράκ σε επίπεδο δηλαδή αυτών που ωφελούνται ε, σκανδάλων, διαφθοράς κτλ η μείωση της ε, έκφρασης βίας στο Ιράκ τον τελευταίο καιρό μπορεί να αποδοθεί στην καλύτερη αστυνόμευση της χώρας ή σε άλλους παράγοντες. Ευχαριστώ κύριε Αρλάκη, ο κύριος Λατσμπέργη σε ένα λεπτό. Ε, ε, η ερώτησή μου αφορά τα Ηνωμένα Έθνη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα σχετικά με το στρατόπεδο Ασράφ και ζήτησε τη σωστή προστασία όλων αυτών οι οποίοι βρίσκονται ουσιαστικά σε πολιορκία. Θεωρούνται υποτίθεται προστατευόμενοι αυτοί οι άνθρωποι. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι γίνεται με αυτή την ψυχολογική βία που υφίστανται, η ψυχολογική τρομοκρατία μέσω των μεγάλων μεγαφώνων, μέσω των ενεργειών βίας, δολοφονιών. Ε, οι Αμερικανοί τους εγκατέλειψαν, οι Ιρακινοί είναι εναντίον τους λέγοντας ότι η παλαιή αλής του φήμης επαναστατική ε, φρουρά θα ξαναρχίσει ε, τρομοκρατικές ε, ενέργειες. Εν πάση περιπτώσει πολύ φοβάμαι ότι θα πέσουμε σε νέες τρομοκρατικές ενέργειες αν δεν υπάρχει προσπάθεια να αποφύγουμε στο μέλλον τραγωδίες τύπου Νταρφούρ ή Σρεμπρένιτσα που θα γελιοποιήσουν ε, για μια ακόμη φορά την οργάνωσή σας και φυσικά τι κάνετε και πώς πιέζετε ε, την Ιρακινή κυβέρνηση και τι συνέπειες θα υποστεί ε, στην περίπτωση που συνεχίσει αυτή την απαράδεκτη υποκρισία την οποία εκφράζει. Μποσκούρτε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζουμε κύριε Μελκάρτ στην Επιτροπή μας από την Ολλανδία. Αναφερθήκατε στο θέμα των χριστιανών, αναφερθήκατε στις εκλογικές διαδικασίες οι οποίες εξελίχθησαν σχετικά καλώς ε, αναφερθήκατε στην δημοκρατία που πρέπει να προστατεύει τις μειονότητες όπως τους χριστιανούς και όλους όσους ε, ε, όπως οι καμπάς που αναγκάστηκαν να φύγουν προς το Ιράν. Τι γίνεται με τη νέα κυβέρνηση, κύριε Μελκόρτ. Τι σχέδια φέρετε να έχει η νέα κυβέρνηση γύρω από τα θέματα αυτά. Τώρα για την κατάσταση ασφαλείας στην χώρα, αυτό συνδέεται όπως ξέρετε και με τους πρόσφυγες στην Ευρώπη. Λέτε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα αλλά όχι όσο καλά θα θέλατε. Ο κύριος Βιντάλ Κουάντρα σε ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ κύριε Μέλκερ για την προσπάθεια την οποία κάνατε και για τον χρόνο που μας αφιερώνετε. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο ε, στην αποστολή σας στο Ιράκ. Ε, ένα θέμα θα ήθελα να θέσω, στο οποίο έχουν αναφερθεί και άλλοι συνάδελφοι. Την κατάσταση δηλαδή στο στρατόπεδο προσφύγων του Ασράφ. Η κατάσταση μέχρι τώρα στο στρατόπεδο Ασράφ, κύριε Μελκέρτη, είναι απαράδεκτη. Ο κόσμος εκεί αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, δεν υπάρχουν ε, ε, τρόφιμα, δεν υπάρχουν φάρμακα, καρκινοπαθείς δεν θεραπεύονται, υπάρχουν ψυχολογικά βασανιστήρια με τις τεράστιες αυτές ε, μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Ε, όλα αυτά φυσικά παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση της χώρας και Ε, μας πληροφορούν κυρία το ότι τις επόμενες μέρες θα μπορούσε να υπάρξει μάλιστα και μία επίθεση χειρότερη από αυτήν η οποία προηγήθηκε τον Ιούλιο όταν σκοτώθηκαν 11 άτομα και αν υπάρξει μια τέτοια άλλη επίθεση τότε πράγματι θα έχουμε να κάνουμε με σφαγή μεγάλου μεγέθους. Γι' αυτό κύριε Μέλκερτ μπορείτε παρακαλώ να δημιουργήσετε μια ομάδα παρατηρητών άμεσα στο στρατόπεδο αυτό κάτω από την αιγίδα των συμμαχικών δυνάμεων γιατί αλλιώς διακινδυνεύεται κύριε Μέλκερτ να υπάρξει πράγματι μια νέα μαζική σφαγή. Μάγερ ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μέλκερταν και δεν μπορεί να με δει εδώ λόγω ακριβώς των, τηλεοπτικών συνεργείων. Εν πάση περιπτώσει κάπως απομακρύνθηκαν. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δίνει για τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών αυτούς τους τελευταίους μήνες έτσι ώστε να μπορέσει ο Νούρι Αλμαλίκη να σχηματίσει την κυβέρνησή του. Και αυτό θα γίνει μέσα Δεκεμβρίου, αν καταλάβαμε. Διαβετώμε λοιπόν αν αυτή η συνταγή λιβανικού τύπου η οποία ακολουθήθηκε για την αντιπροσώπευση των διαφόρων φιλετικών ομάδων στην κυβέρνηση είναι η καταλληλότερη συνταγή για να ξεπεραστούν ή φιλετικές συγκρούσεις ε, και διαφορές. Στα πλαίσια της έκθεσης του Ερυθρού Σταυρού μαθαίνουμε ότι η φιλετικες συγκρουσεις και διαφορες στα πλαισια της εκθεσης του ευθρου σταυρου μαθαινουμε οτι η κατασταση για τον άμαχο πληθυσμό είναι ιδιαίτερα κακή ακόμα. Εξεπλάγει από τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Αλμαλίκη λέγοντας ότι ε, ε, δεν αμφισβητεί τη συμφωνία στην οποία έχει καταλήξει με τις δυνάμεις κατοχής. Έτσι τις χαρακτήρισε. Ποια είναι η άποψή σας κύριε Μέλκερτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τα τελευταία σημεία τα οποία σημειώθηκαν. Δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω Αυτά τα οποία έχει πει ο Πρωθυπουργό Αλμαλίκη είναι δική του αποκλειστικά ευθύνη για τη γενικότερη κατάσταση την ανθρωπιστική. Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση εδώ ανάμεσα σε περιοχές της χώρας. Υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στο βόρειο τμήμα, στην περιοχή του Κουρδιστάν δηλαδή, και σε άλλα τμήματα του Ιράκ, τα οποία είναι σχετικά ασφαλή, αν και συμβαίνουν κάποια πράγματα βέβαια, και κάποιες άλλες περιοχές όπου συμβαίνουν σε καθημερινή, θα έλεγα, βάση προβλήματα, όπως το Μαγκάτ, Μακούμπα και Μοσούλη. Πάντως ο μέσος όρος των βίαιων ενεργειών έχει σαφέστατα μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα μαύρα χρόνια θα έλεγα αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να πει κανείς σήμερα ότι το Ιράκ είναι ένα ανασφαλές μέρος συνολικά, παρόλα αυτά υπάρχουν περιοχές όπου η κατάσταση είναι δύσκολο να περιγραφεί για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τους παλινοστήσαντες. Βλέποντας λοιπόν ποια είναι κατά περίπτωση η κατάσταση αυτών των πληθυσμών είναι ο μοναδικός τρόπος έτσι ώστε να αξιολογήσουμε τις συνθήκες των προσφύγων ε, ε, και των ε, εσωτερικά εκτοπισμένων μέσα στο Ιράκ κατοίκων που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα θα ήθελα να είμαι επιφυλακτικός για τις πιθανές συγκρίσεις των πολιτικών εξελίξεων στο Ιράκ με αυτές στο Λίβανο. Κατάλαβα γιατί τίθεται βέβαια το συγκεκριμένο θέμα, αλλά η φύση των πολιτικών διαδικασιών στο Ιράκ είναι ιδιαίτερη θα έλεγα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κάτι το ξεχωριστό. Επιπλέον βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα πρόορη φάση συνεργασίας επί τη βάση του νέου συντάγματος και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν οι εξελίξεις θα είναι ικανοποιητικές. Μόνο ο χρόνος θα μας φωτίσει. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Βιντάλ Κουάδρας για τις ακούραστες προσπάθειες τις οποίες κάνει για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων. Θα ήθελα επίσης να τον διαβεβαιώσω ότι όλες οι εκθέσεις και όλα τα μηνύματα τα οποία έρχονται από τη δική σας πλευρά και από την πλευρά των συναδέλφων εξετάζονται πάρα πολύ σοβαρά και θεωρούμε ότι είστε μία από τις πηγές για την εποπτεία την οποία προσπαθούμε να ασκήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Ακούγοντας αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λάντσπεργκης θα ήθελα να πω ότι οι δυνατότητες για την γιουνάμι στο Ιράκ επί τη βάση της εντολής μας είναι περιορισμένες καθοδηγούνται φυσικά από τις βασικές αρχές των διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκεί δεν υπάρχουν παραχωρήσεις. Συνεργαζόμαστε με την ύπατη αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει μια πιο προληπτική ευρύτερη εντολή για να αντιμετωπίσει τα θέματα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνεργαζόμαστε στενά με την Ιρακινή κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της χώρας. Το θέμα δεν είναι απλά διεθνών συμβάσεων και στο Ιράκ γίνεται μια συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά και δεν θα με εκπλήξει καθόλου εάν στα πλαίσια του νέου γαλαξία που θα είναι η νέα κυβέρνηση και που θα συσταθεί σε ευρύτερη βάση από ό,τι στο παρελθόν και με ένα κοινοβούλιο Ιρακινό πιο αποφασιστικό, τα θέματα αυτά και στο ίδιο το Ιράκ θα γίνουν αντικείμενο συζήτησης. Νομίζω ότι και εμείς από δική μας πλευράς, από δική μας πλευράς λοιπόν και εμείς θα πρέπει να σεβαστούμε τους Ιρακινούς θεσμούς που θέλουν να ασχοληθούν με όλα αυτά, αλλά και όλοι έχουμε την συλλογική ευθύνη να εργαστούμε σύμφωνα με τις βασικές καθολικές αξίες που εμπνέουν τα Ηνωμένα Έθνη. Γι' αυτό ασκούμε την εποπτεία αυτή η οποία μας καθιστά ικανούς να είμαστε συγκεκριμένοι στην αλληλοεπίδραση την οποία έχουμε με τους Ιρακινούς για αυτά τα οποία βλέπουμε και τι πρέπει να αλλάξει. Αλλά είναι ευθύνη της κυβέρνησης του Ιράκ να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και είναι σημαντικό οι αποφάσεις αυτές να γίνονται αντικείμενο σεβασμού και ταυτόχρονα να είναι συμβατές με τις διεθνώς αποδεκτές αρχές προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις υπόλοιπες ανθρωπιστικές αρχές. Δεν θα μπορούσα να πω τι σκοπεύει να κάνει η νέα κυβέρνηση σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων. Να παρατηρήσω όμως ότι όλοι οι πολιτικοί ηγέτες έχουν συμφωνήσει καταδικάζοντας τις απέσιες επιθέσεις σε κάποιες εκκλησίες τον μήνα Οκτώβριο και υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση εδώ ότι το μέλλον του Ιράκ θα πρέπει να θεμελιωθεί στον σεβασμό για όλους ανεξαρτήτως των φιλετικών ή θρησκευτικών καταβολών τους. Έχουν βέβαια τα τελευταία χρόνια συμβεί πάρα πολλά στο Ιράκ. Δυστυχώς όλα αυτά έχουν λειτουργήσει σαν κίνητρο για αυτούς οι οποίοι θα ήθελαν να υπάρξουν περισσότερο έντονες θρησκευτικές διαφορές και να προωθηθούν συγκεκριμένα φιλετικοθρησκευτικά συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα έχει πλέον διαμορφώσει μια παράδοση στη συγκεκριμένη χώρα. Στο παρελθόν δεν ενδιαφερόμεθα και δεν γνωρίζαμε ποια είναι η καταβολή των συγκεκριμένων πολιτών Τώρα αυτό ορίζεται και ε, συνοδεύει τον κάθε Ιρακινό πολίτη και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις αρχές του Ιράκ να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται με τις εγκαταστάσεις των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικότερα όμως θα πω ότι για όλες αυτές τις οργανώσεις και τα κράτη-μέλη που λειτουργούν στα πλαίσια της διεθνούς ζώνης υπάρχει ανάγκη πάντα για βελτίωση της παρεχόμενης προστασίας. Θεωρούμε ο κίνδυνος να μειωθεί στο μέλλον. Είναι πολύ καλοδεχούμενη η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων Just Lex και θεωρούμε ότι και η νέα κυβέρνηση θα καθορίσει την εσωτερική τάξη και τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου σαν ένα από τα βασικά συστατικά της πολιτικής της που θα καθορίσει το μέλλον της χώρας. Για τις εμπορικές δραστηριότητες. Πολλά εξαρτώνται από τις επενδύσεις στις υποδομές για το πετρέλαιο και την αύξηση παραγωγής πετρελαίου. Υπάρχει επίσης και μία αύξηση στο λεγόμενο real estate και στις τουριστικές δραστηριότητες, αλλά παρόλα αυτά η ε, ποικιλότητα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την Ιρακινή οικονομία είναι κάτι που απασχολεί την κυβέρνηση. Η διεθνής βοήθεια σε σχέση με τη βοήθεια προς το Αφγανιστάν. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Καταρχάς το επίπεδο της διεθνούς βοήθειας για ανθρωπιστικούς λόγους ιδιαίτερα όταν διακρίνει κανείς τη συνεισφορά των Αμερικανών και τις άλλες χώρες, θα δει ότι είναι πολύ μικρότερη η διαφορά από ό,τι στο Αφγανιστάν. Εμείς εκτιμούμε αυτή τη στιγμή τις συνεισφορές μέσω του Ταμείου του Ιράκ για την ανοικοδόμηση και το οποίο είχε στη διάθεσή του τα τελευταία 5-6 χρόνια γύρω στο 1,35 δις δολάρια. Υπάρχουν προβλήματα με την διαφθορά. Ξέρετε ότι στον δείκτη ε, διαφθορά στο Ιράκ είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ε, Παρ' όλα αυτά απαιτούνται επενδύσεις στον τομέα της, ε, του σεβασμού του κράτους δικαίου που θα βελτιώσει την κατάσταση. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, η μείωση των βίαιων δραστηριοτήτων και ο ρόλος των δυνάμεων καταστολής και δυνάμεων ασφαλείας Υπάρχει ανησυχία σχετικά με τις ικανότητες των Ιρακινών δυνάμεων η οποία έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο. Όταν λέω όμως κατά μέσο όρο ε, εννοώ ότι υπάρχουν και ε, διαφορές σχετικά με το είδος της ενασχόλησης, της δραστηριότητας, την περιοχή στην οποία δρούν οι δυνάμεις ασφαλείας. Πολλά μένει να γίνουν και κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης των αστυνομικών δυνάμεων και εδώ η εμπλοκή ορισμένων χωρών μελών που υποστηρίζουν το Ιράκ προς την κατεύθυνση αυτή είναι ένας πολύ καλός μεσοπρόθεσμα τρόπος για την προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάστασης δημιουργίας μιας κανονικής χώρας όπου οι πολίτες μετακινούνται ελεύθερα, οι επενδυτές επενδύουν και η οικονομική ανάκαμψη και η καταπολέμηση της ένδυας θα είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τους πολίτες αύριο. Είμαστε μακράν όμως αυτής της κατάστασης λόγω της ανασφάλειας που σοβεί εκεί. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και πάντα η διεθνή συμμετοχή θα μετατρέψει την αισιοδοξία νομίζω σε πραγματικότητα. Ευχαριστώ κύριε ε, Μέλκερτ. Ο διάλογος που προηγήθηκε ήταν ιδιαίτερα καρποφόρος λόγω της διαθεσιμότητας την οποία επιδείξατε. Θα συνεχίσουμε τις επαφές μας στον τομέα αυτό το συντομότερο δυνατόν. Cari colleghi, oggi ναι, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτηση για τα τελευταία γεγονότα στη Δυτική Σαχάρα. Ακούσαμε ε, τον κύριο Τσαλέκ, τον εκπρόσωπο του μετόπου Πολυσάριο. Τώρα θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φασιφύρη. Ο κύριος Φασιφύρη δέχτηκε την πρόσκληση που του αποστήλαμε. Ε, discutere questo delicato tema. Come ε, lei sa, signor Ministro, <clears throat> il Ο κύριος Φασιφύρη λοιπόν θα αναφερθεί και στο ψήφισμα που υιοθετήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα το θέμα αυτό προκάλεσε κάποια αμηχανία στη χώρα του. Θα ήθελα να διευκρινίσω εδώ ότι το ψήφισμα αυτό ε, δεν ήταν θα έλεγα καθρέφτης μία συγκεκριμένης αθνικής αντιπροσωπείας αλλά ήταν αντικείμενο και καρπός διαβούλευσης όλων των πολιτικών ομάδων ανεξαρτήτως εθνικών ε, καταγωγών. Λοιπόν, ε, προσπαθώ να εκπροσωπήσω το σύνολο λοιπόν του Κοινοβουλίου. Είχα τη δυνατότητα κατηδία να το πω. Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για τις απώλειες ανθρώπινης ζωής οι οποίες προκλήθηκαν από τα συμβάντα τα οποία είναι αντικείμενο και τη σημερινή συζήτηση. Σε ό,τι σας αφορά κύριε Υπουργέ θα ήθελα να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας και για τις οικογένειες των ε, θυμάτων ε, των ε, δυνάμεων ασφαλείας του Μαρόκου. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μην ξεπεράσετε παρακαλώ τα 10 λεπτά και να είστε πλήρης όμως και συνεκτικός. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και περιμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψε μαζί σας. Και ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ε, για την ευγενική πρόσκληση. Με καλέσατε για να συζητήσουμε, να σας ακούσω, να απαντήσω και να σημειώσω τα σχόλια της παρατηρήσεως, ε, την ανάλυση της κατάστασης για το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Και θα ήθελα να τηρήσω το χρόνο μου. Καταρχήν θα ήθελα να επιβεβαιώσω για μια ακόμη φορά την δέσμευση του Μαρόκου να αναπτύξει και να εμβαθύνει τη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια στρατηγική που εφαρμόσαμε μέσα μετά την ανάκτηση της ανεξαρτησίας μας και καλύπτει όλο το πολιτικό φάσμα του πολιτικού βίου του Μαρόκου. Και μάλιστα αυτή η δέσμευση είναι μονοσήμαντη, γιατί όσο πλησιάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνουμε ότι έχουμε στερνιζόμαστε τις αξίες και τις αρχές και όσο περισσότερο συμμεριζόμαστε αυτές τις αξίες και τις αρχές και τις διατάξεις τόσο θα προοδεύουμε και εμείς. Εμείς δεν αρνούμαστε την αμοιβαία ανάμειξη και συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Γειτονία, έχουμε διαδοχικά σχέδια εργασίας, έχουμε τη συζήτηση για το προηγμένο καθεστώς. Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε τις δεσμεύσει μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θεωρούμε ότι η πολιτική γειτονία είναι παρέμβαση στις εξωτερικές μας υποθέσεις. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι δίνουμε νέα πνοή στον πολιτικό μας βίο και μία όθηση για πρόοδο. Το προηγμένο καθεστώ ε, που δόθηκε στο Μαρόκο έγινε δεκτό και είναι πρόσδεκτο στο Μαρόκο και τίνει προς μια και κανονιστική σύγκληση, γιατί την πολιτική σύγκληση την έχουμε διατρανώσει. Είμαστε υπέρ της ε, διατήρησης της ειρήνης. Είμαστε η μόνη χώρα του Νότου που συμμετέχει στην επιχείρηση Alter για την αποκατάσταση ειρήνης στη Βοσνία Ζεγοβίνη και είμαστε η πρώτη ε, χώρα που έχει υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε η μόνη χώρα του Νότου που έχει τέτοια ομάδα με μεικτή ε, συμμετοχή, με συμμετοχή όχι μόνο κυβερνητικών αλλά και εκπροσώπων ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι άπειρα τα παραδείγματα που δείχνουν πώς εξυγχρονίζεται, προοδεύει, μεταμορφώνεται το Μαρόκο και αναπτύσσει αυτές τις ειδικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που αντιμετωπίζει ορισμένες δυσκολίες στην περιοχή, στο Μαγκρέμπ. Εκεί είμαστε οι χειρότεροι μαθητές της επιδόσης ό,τι αφορά την αφρικανική ολοκλήρωση. Έχουμε κλειστά σύνορα με τους αλγερινούς γειτονές μας, σύνορα που μένουν κλειστά για αδιαφανείς λόγους που πραγματικά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και άλλα ζητήματα σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Σε ό,τι αφορά και το Έχεις Περιβάλλον. Έχουμε προβλήματα στη Δυτική Σαχάρα. Έχαμε πολύ λεπτές εξελίξεις στη Μαυριτανία, Μαλή, Νιγηρία, Γκάμπια, Γουινέα Μπισάου. Και αυτές οι εξελίξεις ε, μας προβληματίζουν και από στρατηγική άποψη. Τώρα, το θέμα της ε, Σαχάρας. Έχω σχετική τεκμηρίωση για το θέμα αυτό για όποιον ενδιαφέρεται, με κάποιες ιστορικές αναφορές και με απάντηση σε πολύ συχνές ερωτήσεις. Γι' αυτό και δεν θα ήθελα να επεκταθώ στο θέμα αυτό. Το Μαρόκο πέρασε μια ιδιάζουσα φάση απεικιοποίησης, μεικτή, ε, γαλλική στο κέντρο και στο βορρά και νότο ισπανική. Και σε αυτό το φαινόμενο της ε, αποαπικιοποίησης και της ανάκτησης της πλήρους κυριαρχίας ε, περάσαμε αυτή τη διαδικασία με διάφορες φάσεις. Και σε ό,τι φορά την ε, ζώνη της Σαχάρας, που δεν περιλαμβάνει τη Δυτική Σαχάρα, αλλά είχαμε και άλλες ζώνες υπό Ισπανική κατοχή που ανακτήσαμε, γιατί ήταν δικές μας. Είχαμε το 58 τη ζώνη Ταρφάγια σε συμφωνία με την Ισπανία, το Συνδιεφνή το 69 και τη συμφωνία της Μαδρίτης το 75 για την Δυτική Σαχάρα. Το 1965 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε από την Ισπανία να διαπραγματευτεί με το Μαρόκο την ε, ε, επιστροφή του στη και της Δυτικής Σαχάρας. Αυτή, αυτό ήταν ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης. Το Ισπανικό Καθεστώ τότε προτίμησε να γίνει σε δύο φάσεις. Η ζώνη συντηφινή επιστράφει, επιστράφει το 69, αλλά ήταν κάπως αργά πια γιατί είχε αλλάξει στο μεταξύ το διεθνές προσκήνιο και οι εξελίξεις στο Μαγκρέπ το ίδιο. Εξού και ξεκίνησε αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ Αλγερίας και Μαρόκου για το θέμα της Σαχάρας. Το Πολυσάριο δεν υπήρχε, το μέτωπο Πολυσάριο δεν υπήρχε κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Απικιοκρατίας. Το Πολυσάριο γεννήθηκε, ιδρύθηκε χάρη σε μία πρωτοβουλία του Λιβικού καθεστώτος που υποστήριξε εκεί η Αλγερία στο συγκεκριμένο ειδικό πλαίσιο. Το μέτωπο Πολυσάριο δεν είναι ο μοναδικός και θεμητός εκπρόσωπος του λαού της Δυτικής Σαχάρας, των Σαχαροϊτών. Δεν κατοχυρώνεται κάτι τέτοιο σε κανένα έγγραφο το ΙΕ. Δεν έχει ούτε λαϊκή βάση, ούτε νομικό καθεστώς, ούτε οποιαδήποτε δημοκρατική έκφραση που να νομιμοποιούν το Πολυσάριο ως εκπρόσωπο των Σαχαροϊτών. Η μεγάλη πλειοψηφία των Σαχαροϊτών ε, θεωρούν ότι είναι Μαροκινοί και ζουν αυτή την μαροκινότητά τους σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Ούτε για τον ΟΗΕ είναι εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο το Πολυσάριο. Στι διαπραγματεύσει όμω με το Μαρόκο έχει πρωταγωνιστική θέση και προσπαθούμε να βρούμε μαζί με το Πολυσάριο μια οριστική λύση σε αυτό το θέμα. Το Μαρόκο θεώρησε καθήκον του να δώσει μια απάντηση στην έκκληση του 2004 όταν ο ΙΕ ζήτησε από τα εμπλεκόμενα μέρη να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις. Σε αυτή την, σε αυτή την έκκληση ανταποκρίθηκε το Μαρόκο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί προτείναμε μία λύση με βάση μία απλή πρωτοβουλία που δεν ήταν κλειστή στη διαπραγμάτευση, συνάδει με το διεθνές δίκαιο, με τη διεθνή νομιμότητα, ως συμβιβαστική λύση και ως ρεαλιστική απόπειρα αναζήτησης μιας ευκταίας πολιτικής λύσης. Από τότε που καταθέσαμε αυτή την πρόταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το Συμβούλιο Ασφαλείας τη δέχτηκε ως αξιόπιστη και σοβαρή προσπάθεια εκ μέρους του Μαρόκου, κάτι που επιβεβαιώνει την νομιμότητα και το θεμητό χαρακτήρα αυτής της διαδικασίας, που δυστυχώς όμως από την αρχή της κιόλα καταρρίφθηκε για παράδειγμα, ο Αλγερινός ε, πρόεδρος είπε ότι ήταν ε, από την αρχή καταδικασμένη σε θάνατο και ότι η κυριαρχία, το Μαρόκο θεωρούσε ότι είχε κυριαρχία στην περιοχή. Ήταν πολύ σαθρά αυτά τα επιχειρήματα και άλλωστε είχαν αφισβητηθεί και από τον ΟΗΕ. Από τότε που καταθέσαμε αυτή την πρόταση, που είχε φανεί ότι ε, λάμβανε και την ε, διεθνή υποστήριξη, υιοθετήσαμε και στο Μαρόκο μία στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική ήταν σαφής. Ήδη από το 2007 στηρίζεται σε τρία είδη δράσεων. Η πρώτη ήταν ε, μία έκκληση να ενθαρρύνουμε με προγραμματισμένες δράσεις τα θέματα της ε, καταστρατήγης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαχάρα. Δεύτερον, ε, αυτή την υποτιθέμενη ε, μίξου εξουδιωτημένη χρήση των, του πλούτου της Σαχάρας και τρίτον να πει ότι η Σαχάρα είναι μια, ένα κράτος που βρίσκεται υποκατοχή από το Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, αυτή η τρίτη άξονη είναι μια στρατηγική που ξεκίνησε από το 2007 και ήταν μια προπαγάνδα ουσιαστικά που κινητοποιήθηκε ε, εις βάρος, και που ακούγεται, εις μας και που ακούγεται σε πολλές περιοχές και από πολλές φωνές. Τώρα, τι συνέβη στο Λαγιούν. Καταρχήν, υπάρχει το θέμα της υπερηφάνειας. Είμαστε υπερήφανοι που μας επέτρεψαν, που επιτρέψαμε με κάθε ελευθερία να κατασκευαστούν τέτοιοι καταβλισμοί. Αισθάνομαστε υπερήφανοι που αντί να κλείσουμε αυτό το καταβλισμό όταν το Πολυσάριο έλεγε ότι ήταν κλειστός, εμείς τον αφήσαμε ανοιχτό, Γιατί υπήρχε ένα είδος αποκλεισμού από φάρμακα και τρόφιμα. Εκεί 600.000 αυτοκίνητα μπενόβγαιναν κάθε μέρα. Μάλλον όχι, 600 με 1.000 αυτοκίνητα μπενόβγαιναν κάθε μέρα, σε αντίθεση με τα επιχειρήματα του Πολυσάριου και της Αλγερίας. Ο καταβλισμός ε, διαλύθηκε με ειρηνικό τρόπο και δεν νομίζω ότι σε καμία δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα θα ήταν τόσο ειρηνική αυτή η διάλυση. Και μάλιστα τα θύματα βρίσκονται στην πλευρά των στρατιωτικών δυνάμεων του Μαρόκου. Δεν υπήρχε ούτε ένα θύμα αμαχοπληθισμού παρόλο που πολλοί ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκαναν λόγο για γενοκτονία και εθνοκάθαρση. Μάλιστα σήμερα η επιχείρηση αυτή ολοκληρώθηκε και είναι επιβεβαιωμένο ότι δεν υπήρξε καμία βία εκ μέρους μας. Εμείς ήμασταν τα θύματα της βίας. Η αστυνομία αντιμετώπισε βόμβες κοκτέιλ μολότοφ, αντιμετώπισε εγκληματίες που προσπάθησαν να την κατασφάξουν ήταν άδικες οι κατηγορίες που ακούστηκαν. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, γιατί μου επισημαίνει ο Πρόεδρος ότι έχω ξεπεράσει το δεκάλεπτό μου. Είμαι στη διάθεσή σας πάντως για να διαλευκάνω στο μέτρο του δυνατού τις απορίες σας. Σας ευχαριστώ. 20 ζήτησαν το λόγο στον ελάχιστο χρόνο που μας έχει μείνει στη διάθεσή μας και δυστυχώς θα πρέπει να σας περιορίσω, να περιορίσω την κάθε παρέμβαση σε ένα λεπτό το πολύ. Ο κύριος Αλαφράγκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό του Μαρόκου εκ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Χαρακτηρίσατε ως εσπευσμένο και άδικο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Υπουργέ. Πολλά όμω ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούν ε, άδικο και σπευσμένο τον τρόπο με τον οποίο το Μαρόκο διέλυσε τον καταβλισμό του Ισλαγιούν. Σε μια, σε μια συνέντευξη στην ΠΑΗΣ ε, της Κυριακής 28ης ε, Νοεμβρίου είπατε, δηλώσετε κύριε Υπουργέ ότι δεν βασανίσατε κανέναν, άδι, ε, κανέναν αθώο. Δηλαδή οι μία αθώοι μπορεί να βασανίστηκαν. Μπορείτε να μας ευκρινίσετε αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις ακρότητες. Η ειδική ανταποκρίτρια του Ελμούντο απελάθη από το Μαρόκο, ενώ στο τελευταίο της άρθρο είπε ότι από τις 130 κρατούμενους Σαχαραουίτες, ένας κατηγγείλει ότι το πενταήμερο που ε, είχαν, είχαν δηλωθεί ως εξασφανισμένοι, είχαν υποστεί βιασμό με φιάλες και τους υποχρέωσαν να πιούν τα ίδια τους τα ούρα μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι στα πλαίσια της ε, συμφωνίας εταιρικής σχέσης ε, που έχουμε ε, δικαιούστε να απελάβνετε έναν δημοσιογράφο όταν διαφωνείτε με το περιεχόμενο του άρθρου που συνέταξε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ, είναι ένα κυρίαρχο θεσμικό όργανο και είναι κυρίαρχο των αποφάσεών του και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών που μας εξέλεξαν και που είναι υπέρ των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη ελευθερία έκφραση και τη ελευθεροτυπίας. Αυτέ οι αξίε βρίσκονται και στην καρδιά τη ε, στρατηγική συμφωνία σύνδεση ε, με το Μαρόκο και δεν ε, δυνάμεθα ούτε οφείλουμε ούτε μπορούμε να παραγνωρίσουμε όλες αυτές τις αξίες. Η κυρία Γκόμες, ένα λεπτό. Κύριε Υπουργέ, μάλλον κύριε Υπουργέ στα γαλλικά. Θεωρούμε ότι το Μαρόκο είναι υπόλογο για τις κρατήσεις, τους τραυματισμούς, τους θανάτους, αυτούς που εξαφανίστηκαν μάλλον κατά τη διάρκεια των τελευταίων συμβάντων στον καταβλισμό. Σύμφωνα με δυτικούς ε, πόρους ε, πληροφόρησης, ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ανάμεσα σε 500 με 600 θα ήθελα να σας ζητήσουμε λοιπόν να επιτρέψετε την είσοδο στο Αγιούν των μελών του Κοινοβουλίου και του τύπου. Θέλω να με διαβεβαιώσετε ότι εγώ ίδια τις επόμενες εβδομάδες θα πάω στο Αγιούν να μιλήσω αλεύθερα με τους κατοίκους και να συλλέξω τις πληροφορίες που χρειάζονται. Ε, εσείς είσαστε υποτίθετε σε διαπραγματεύσεις με το μέτωπο Πολυσάριο στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών γιατί προσπαθήσατε εδώ να πείτε ότι ο συνομιλητής σας στο μέτωπο Πολυσάριο ε, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Κυρία Νέιτς, ένα λεπτό. Κύριε Υπουργέ, η πολιτική μου ομάδα έχει συνυπογράψει το κοινό ψήφισμα το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν συμφωνώ με όλα όσα λέγονται στο ψήφισμα αυτό αλλά πρόκειται για ένα επίσημο κείμενο ενός κυρίαρχου πολιτικού οργάνου. Και φυσικά έχετε το δικαίωμα να έχετε τη δική σας άποψη γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ όμως ότι η νομιμότητα του συγκεκριμένου εγγράφου είναι και αυτή δεδομένη. Επί της ουσίας τώρα. Λέγεται ότι το συγκεκριμένο αυτό ο συγκεκριμένος καταβλισμός έξω από το Αγιούν ε, το έκαναν αυτό για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Ήθελαν θέσεις εργασίας, ήθελαν ε, ε μικρές εκτάσεις ε, γης για να καλλιεργήσουν και κάτι τέτοιο τους το είχαν υποτίθεται υποσχεθεί. Ταυτόχρονα μας λέτε και δεν αμφιβάλλω για την αλήθεια ότι η περιοχή του Αγιούν αναπτύχθηκε οικονομικά τον τελευταίο καιρό με πολύ μεγα, υψηλούς ρυθμούς. Πώς ε, λοιπόν ε, εδώ συνδυάζεται, εξηγείται αυτή την ασυμβατότητα ανάμεσα στο ρυθμό ανάπτυξης και τα προβλήματα των κατοίκων. Ρωμέβα, ένα λεπτό. Κύριε, Κύριε Υπουργέ, εν συντομία, με σόκαρε το σχόλιο σας για το ότι δεν διέπραξε βιότητες τα μέλη των, το μαροκινών δυνάμεων. Και πού, πού βρίσκονται το τι εξαφανιστέντες, μπορείτε να μας πείτε. Άλλωστε, ε, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι ψήφισμα του ΕΛΚ, αλλά κοινό ψήφισμα όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφού υποτίθεται ότι κόπτεστε για την διεθνή νομιμότητα, γιατί δεν επιτρέπετε τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στη Δυτική Σαχάρα. Και αν δεν έχετε τίποτα να κρύψετε, γιατί εμποδίζετε τους παρατηρητές να κάνουν το έργο τους τους α, όσους θέλουν να, προσ να επισκεφθούν την, τον καταβλισμό. Και γιατί εκμεταλλεύεστε τους φυσικούς πόρους α, ε, μιας που δεν σας ανήκει, όπως είναι η Δυτική Σαχάρα. Ο κύριος Μέγερ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, εσείς ως δύναμη, παράνομη δύναμη κατοχής της μη αυτόνομης περιοχής της Δυτικής Σαχάρας, γιατί έτσι αποκαλείται στο Διεθνές Δίκαιο αυτή η ζώνη, είπατε ότι αποφασίσατε μάλλον ότι δεν θέλετε μάρτυρες στην ε, ζώνη αυτή. Γι' αυτό απαγορεύεται την ε, ελεύθερη κυκλοφορία βουλευτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και οποιοδήποτε, οποιοδήποτε διεθνού παρατηρητή μέσω μαζικής ενημέρωσης δεν θέλετε μάρτυρες ε, σε αυτές τις εγκληματικές ενέργειες που διαπράτεται στην Δυτική Σαχάρα εσείς και οι μαροκινές στρατιωτικές δυνάμεις. Εγώ σας ζητώ να εφαρμόσετε τη διεθνή νομιμότητα και το τελευταίο ψήφισμα ε, για το δεύτερο σχέδιο Baker που εγκρίθηκε ομόφωνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα πρέπει αυτό το σχέδιο να εφαρμοστεί και να απελευθερώσετε όλους τους παράνομα ε, κρατούμενους, παράνομα πολιτικούς κρατούμενους. Και ως παράνομη δύναμη κατοχής ε, θα ήθελα να ζητήσω από το Μαρόκο να σεβαστεί και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Ο κύριος Μιγιάν Μόν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που ε, διευκρινίσαμε τον οριζόντιο και τον κοινό χαρακτήρα του ψηφίσματος της περασμένης εβδομάδας. Είναι συνενωτικό το ψήφισμα. Θα ήθελα να υποβάλω τις ε, δύο ερωτήσεις που έθεσα και στον εκπρόσωπο του μετόπου Πολυσάριο. Γιατί δεν κατέστη δυνατή διάλυση του, του καταβλισμού, γιατί είπατε ότι είχατε ειρηνικές ε, διαβουλεύσεις με τους διοργανωτές της διαδήλωσης και μάλιστα είχαν ε, ξεκινήσει και πάλι η συνομιλία στη Νέα Υόρκη. Πού οφείλεται αυτή η παρεκτροπή και πώς βλέπετε τις προοπτικές των νέων συνομιλιών που ξεκίνησαν στη Νέα Υόρκη. Τι προβλέψεις κάνετε για την έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ κύριο Σπαρνιό για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Είναι κρίσιμη αυτή η στιγμή που έρχεσαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε να έρθει και ο Αλγερινός Υπουργός Εξωτερικών, βέβαια έστειλε επιστολή από ό,τι ξέρω στον Πρόεδρό μας. Θα ήθελα να σας θέσω μία ερώτηση μόνο. Είπατε πριν από λίγο ότι η συμβαστική λύση που προτείνεται το 2004 έγινε δεκτή λήφθη υπόψη από τα Ηνωμένα Έθνη και πρόσφατα ο Κρίστοφα Ρώσο, ειδικός εντεταλμένος του Γενικού Γραμματέα, έκρινε δίκη και σοβαρή την πρόταση αυτονομίας που πρότεινε το Μαρόκο για τη Δυτική Σαχάρα. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόσφατα επαραλήθηκαν οι διαπραγματεύσεις στον ΟΗΕ για το θέμα αυτό, προκειμένου να προωθηθεί το σχέδιο για την αυτονομία της Δυτικής Σαχάρας. Δεύτερη ερώτηση και ολοκληρώνω. Γιατί είχαμε αυτά τα επεισόδια σήμερα, αυτή τη στιγμή ειδικά, δηλαδή τη στιγμή της έναρξης ή της επανάληψης των διαπραγματεύσεων. Πού οφείλεται αυτή η σύμπτωση, μπορείτε να μας εξηγήσετε. Ο κύριος Βάγκλη, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ακούσαμε δύο αντιφατικές ε, παρουσιάσει του προβλήματος της ε, ε, Δυτικής Σαχάρας σήμερα. Δεν θέλω να προτρέξω. Οι εμπειρογνώμονες μεταξύ των διπλωματών μπορούν πολύ πιο καλύτερα να εκτιμήσουν τα πράγματα και να τα παρουσιάσουν και πέρα στο Υπουργείο Εξωτερικών του Μαρόκου. Νομίζω ότι η αντίδραση δεν ήταν σωστή και ότι προσπαθείτε να βρείτε επίσης και ε, κάτι να μας προσάψετε εμείς που υπογράψαμε αυτό το ψήφισμα. Γιατί πιστεύετε ότι το Μαρόκο που είναι ένα δημοκρατικό κράτος και εταίρος μας μπορεί να αγνοεί ψηφίσματα του ΙΕ. Θα συμφωνούσατε να ορίσουμε έναν έκτακτο απεσταλμένο για τη Δυτική Σαχάρα που να συνεργαστείτε μαζί του ο κύριος ένα λεπτό. Η κυρία ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα θέματα. Ο Ισπανός ε, συνάδελφος κύριος Μάιερ, μέλος της Επιτροπής αυτή, ήθελε αρχές, αρχές ε, Νοεμβρίου με δημοσιογράφους να πάει στο Αλαγιούμ για να δημιουργήσει μια εικόνα του ανήθηκε όμως η αστυνομία του Μαρόκο την ε, του εκεί όπως και ε, ο κύριος ε, Μακταλέν που από την Γερμανική Βουλή που θέλησε να πάει εκεί και που έτυχε πραγματικά ε, πολύ κακής μεταχείρισης και δεν του επιτράπηκε η, η, η μετάβασή του εκεί. Θα ήθελα να ξέρω γιατί το εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του κυρίου Μάγερ δεν το επιτράπηκε να πάει στη Δυτική Σαχάρα. Απαντήστε μου παρακαλώ. Η δική μου πολιτική ομάδα και θεωρεί ότι η κατοχή της Δυτικής Σαχάρας και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων εκεί ε, είναι ο λόγος για τον οποίο ε, έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Εδώ και πολλά χρόνια αγνοεί το Μαρόκο το ψήφισμα του ΟΗΕ για ένα δημοψήφισμα. Ε, τι θα λέγατε να γίνει αυτό κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Τότε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σήμερα. Εξεπλάγει, όπως και πολλοί από τους βουλευτές, που η ψηφοφορία του ψηφίσματος προβλέπεται για το Δεκέμβριο έχει τώρα οριστεί για τον, ε, ορίστηκε για τον Νοέμβριο, πράγμα που δεν πέτρεπε σωστή ενημέρωση. Βέβαια, Πρέπει επίση να σεβόσαστε τις συζητήσει που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα αποτελέσματα, τα ψηφίσματα. Θα ήθελα να σας πω ότι η ψηφοφορία του ψηφίσματος αυτό το είδαμε όπως έγινε και για τη Γαλλία ε, με το ψήφισμα για τους Ρωμά όπου η Γαλλία αρτήθηκε κατόπιν ε, τα αποτελέσματα του ψηφίσματος. Πρέπει λοιπόν να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη ψηφοφορία για τα ψηφίσματα αυτά. Κατόπιν, το σχέδιο αυτονομίας που προτείνει το Μαρόκο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσει ε, αυτοδιάθεσης που έχουν οι Σαραούι και επίσης γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η έντονη βία κατά των αστυνομικών του Μαρόκο και αυτό σχετίζεται με τη δηλώση του Πολυσάριο. Ευχαριστώ κύριε Αντατή. Ο κύριος Υπουργός το λόγο να απαντήσει. Je remercie, mesdames et messieurs les députés, pour Ευχαριστώ τους βουλευτές για τις ερωτήσεις του. Θα ήθελα να πω ότι χρησιμοποιήθηκαν κάποιες λέξεις με μια πάρα πολύ υψηλή ελαφρότητα θα έλεγα ε, άγνωστη με τη διεθνή νομιμότητα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Άκουσα από εσά να χρησιμοποιείτε τον όρο κατοχή. Βρείτε εσείς σε ένα ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών τη λέξη κατοχή. Λοιπόν, σας προκαλώ να βρείτε στις νομικές υπηρεσίες των Συμβούλων των Ηνωμένων Εθνών τη λέξη κατοχή. Μη χρησιμοποιείτε παρακαλώ τόσο πρόχειρα τις λέξεις αυτές επαναλαμβάνοντας μια προπαγανδιστική πρακτική άλλων. Λέτε ότι το Μαρόκο δεν υπακούει στα διεθνή νομιμότητα και λέτε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος. Εντελώς λάθος. Σας προκαλώ να μου πείτε σε ποια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπάρχει η λέξη από το 2004 για δημοψήφισμα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη και τις γειτονικές χώρες μεταξύ των οποίων και την Αλγερία να συνεργαστούν μεταξύ τους, Μαρόκο, Αλγερία ανάμεσα σε άλλους, για να βρεθεί μία διαπραγματευόμενη ε, ε αμοιβαίως αποδεκτή λύση η οποία αναλαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες που έκανε το Μαρόκο το 2006. Έτσι λέει το Συμβούλιο Ασφαλείας, που να βασίζεται στην αίσθηση του συμβιβασμού και στον ρεαλισμό, έτσι ώστε να υπάρξει αυτοδιάθεση. Μην συγχαίεται το δημοψήφισμα με την αυτοδιάθεση. Το δημοψήφισμα είναι ένας μηχανισμός Ακούω κάποια χαμόγελα σαρκαστικά, αλλά θα ήθελα να μου απαντήσετε. Δεν υπάρχει η λέξη δημοψήφισμα από το 2004 στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Προσπαθήσαμε από το 89 μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 προσπαθήσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν είναι πανάκια, δεν γίνεται. Είναι ένας μειοψηφικός μηχανισμός. Τρία δημοψηφίσματα έχουν γίνει υπό την γίδα των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση 64 συνολικά περιπτώσεων. Ποιος επιβάλλει συνθήκες σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ποιος λέει ότι απαιτώ η λύση να βρεθεί μόνο από ε, δημοψήφισμα και μένει στη θέση αυτό και σε σχέση με το ρόλο της διεθνούς κοινότητας και σε σχέση με το ε, Συμβούλιο Ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε τη λέξη κατοχή, διότι είστε εντελώς εκτός της διεθνούς νομιμότητας και της νομικής ασφάλειας. Εκμετάλλευση φυσικών πόρων τώρα. Έτσι, μιλάτε για εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Αντιστρέφετε την πραγματικότητα. Η Σαχάρα είναι μια φτωχή περιοχή. Η Σαχάρα δεν έχει φυσικούς πόρους που θα επέτρεπαν ε, την εκμετάλλευσή τους για τον τοπικό πληθυσμό. Ε, βοηθιέται από την διεθνή κοινότητα. Δεν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις των φυσικών πόρων. Υπάρχουν οι, τα φωσφορούχα κοιτάσματα μπόχρα που αντιπροσωπεύει το 1% ε, των δραστηριοτήτων των αντίστοιχων στο Μαρόκο και που μένουν σε δραστηριότητα για κοινωνικούς λόγους. Σχετικά με την αλληλεία τώρα, Εκεί μιλάμε για μια δημόσια επένδυση για τις ιδιωτικές επενδύσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη των αλλιευτικών δραστηριοτήτων στον Νότο. Τώρα, το να μην ασχολούμεθα καθόλου με τους φυσικούς πόρους γιατί πρέπει να εκφραστεί το σύνολο του πληθυσμού. Τι θέλετε, θέλετε να τιμωρήσετε τους πληθυσμούς αυτούς. Θέλετε να περιμένετε ένα δημοψήφισμα για να διαβουλευτείτε με τον πληθυσμό αν οι φυσικοί αυτοί πόροι τους ενδιαφέρουν. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, όταν ακούω να μου λέτε ότι υπήρξαν ίσως 500 νεκροί, ενώ όλος ο κόσμος, μα όλος ο κόσμος, μεταξύ των οποίων και το Human Rights Watch και η Amnesty International και η Διεθνής ε, Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πράγματι, εσείς δεν θελήσατε να ανταλάβετε υπόψη σας όλα αυτά βέβαια στο ψήφισμά σας. Το Human Rights Watch είπε ότι δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός. Και εσείς είπατε ότι υπήρξαν 500 ε, και 600 που έχουν εξαφανιστεί. Εγώ ζήτησα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Πολυσάριο να μου δώσουν ονόματα. Δύο, δύο ονόματα μου δώσανε. Και αυτά τα δύο ονόματα είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εν ζωή και έδωσαν τη μαρτυρία τους. Δύο ονόματα μου έδωσαν και είναι εν ζωή και έδωσαν τη μαρτυρία τους και έκαναν και μήνυση μάλιστα διότι θεωρούν ότι τους έχουν βλάψει. Λοιπόν, σιωπούμε σε σχέση με όλες αυτές τις υπερβολές που ακούστηκαν σε σχέση με τη διάλυση του καταβλισμού ότι αρνηθήκαμε να δώσουμε νερό, τρόφιμα και φάρμακα, ότι υπήρξε καταστολή, ότι υπήρξε μαζική σφαγή, ότι υπήρξε αντίσταση απέναντι στην τρομοκρατία. Ενώ ε, το καταβλισμός αυτός ήταν ανοιχτός, όποιος ήθελε έμπαινε, όποιος ήθελε έβγαινε. Μία ανθρωπιστική τραγωδία λέει συνέβη εκεί υπήρχαν αντίστοιχα Auschwitz. Το, το Πολυσάριο χρησιμοποίησε τον όρο Auschwitz για να χαρακτηρίσει αυτό τον καταβλισμό. ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας 20.000 κατοίκων. Κανένας νεκρός παρακαλώ, έχετε την ευγένεια να δεχτείτε την πραγματικότητα. Οκτώ νεκροί εκ των οποίων ένα παιδί 7 ετών. Ζητήσαμε ονόματα για αυτούς όλους τους νεκρούς και δεν μας έδωσε κανένας κανένα όνομα. Όλα αυτά μας παραπέμπει στον Αουγούστο Πινοσέτ υποτίθεται. Λοιπόν, έτσι εσείς αμείβετε τον διάλογο, χαρακτηρίζετε αυτούς που συμμετέχουν. Λοιπόν, αν έχετε ένα νεκρό να μου τον δώσετε και υπήρξαν επτά προπαγανδιστικές ενέργειες. Και αυτή μάλλον η προπαγανδιστική ενέργεια αναφέρεται εδώ σε μαζικές απαγωγές, σε βασανιστήρια. Τώρα ξεχάσαμε τη διάλυση του καταβλισμού και συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στις υποτιθέμενες συλλήψεις και ανακρίσεις στους αστυνομικούς σταθμούς. Είχαν μιλήσει πριν από τη διάλυση του καταβλισμού σε στρατιωτικές <coughs> επιθέσεις. Αυτό είναι λάθος. Είδατε τις ταινίε, είδατε την πραγματικότητα. Οι, στασέρε, οι δυνάμεις ασφαλείας της χωροφυλακής προχώρησαν και αντιμετώπισαν βόμβες, μαχαίρια και όπλα. Αν θέλετε να αρνηθείτε την πραγματικότητα δικαίωμά σα Και ταυτόχρονα ταυτόχρονα προσπαθούμε να συλλέξουμε μαρτυρίες. Ψάχνουμε να βρούμε παιδιά από τη Γάζα για να πούμε ναι βλέπουμε εδώ μία κυρία στη Μαδρίτη η οποία κλαίει γιατί αναγνώρισε το παιδί της. Αλλά αυτά έγιναν στο, στη Γάζα το 2005. parce que les gens sont à la recherche de cadavres. Λοιπόν, αναζητούν πτώματα. Ε, τι αναζητείτε πτώματα, δεν υπάρχουν. Ε, παίρνει ε, τη φωτογραφία ενός εγκλήματος τραγικού που έγινε στην Καζαμπλάνκα το 2005 και ε, πραγματικά εδώ μας δείχνουν νεκρούς. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Αυτά όλα δεν είναι μια εργαλειοποίηση πολιτικών θέσεων για λόγους διαφημιστικούς που προωθούν ορισμένες οργανώσεις και μη κυβερνητικέ κυρίω. Το Πολυσάριο ανάμεσα στο 76 και το 85 δολοφόνησε, σκότωσε ε, Ισπανούς αλληλείς. Όταν ε, η Ένωση των Νέων εκατοντάδων νεκρών, τον, η Ένωση των Συγγενών των νεκρών διαμαρτυρήθηκε. Ε, τι έγινε για όλους αυτούς, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αν ανάμεσά σας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ήδη αποφασίσει ότι η Σαχάρα είναι ανεξάρτητο κράτος, ότι υπάρχει φυλή των Σαχαραουή και ότι το Πολυσάριο τους εκπροσωπεί, τότε δεν έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ένα μόνο λεπτό, Πρόεδρε, για να μου δώσετε τη δυνατότητα να σχολιάσω το ψήφισμα το οποίο θεωρήσατε σωστό να υιοθετήσετε. Δέχεστε να σχολιάσω εγώ σαν εταίρος σας ε, στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου το ψήφισμά σας. Μου το επιτρέπετε. Λέμε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα αποσιωπά πολλές μορφές πραγματικότητας. Δεν αναφέρεται στην παρουσία αξιόπιστων μη κυβερνητικών διεθνών οργανώσεων, που είναι επιτόπου κάποιοι από τους συντάκτες του ψηφίσματος δεν αποδέχθηκαν τα ονόματα Human Rights Watch, Amnesty International και Διεθνής Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δεν συμπεριλάβατε το ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις του Μαρόκου, κυρίως αυτές, ε, δίδουν πληροφορίες γιατί θέλουμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στη χώρα μου. Είναι αξιόπιστες ε, ε, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και τις αγνοείται πλήρως. Αγνοείται επίσης την παρουσία των δημοσιογράφων. Ήταν παρόντες οι δημοσιογράφοι και αναφέρθηκαν άλλωστε. Και τέλος δεν αναφερθήκατε, αν κατάλαβα καλά, και μιας και αναφέρετε το ψήφισμά σας στα ανθρώπινα δικαιώματα του, των Σαχαραουή, οι Μαροκινοί θα ήθελαν να αναγνωρίσετε να αναγνωρίσετε, να αναφερθείτε στο μαρτύριο που έζησαν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν στην διάλυση του συγκεκριμένου καταβλισμού. Δεν δώσατε πληροφορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διερωτάστε ε, για την κατάσταση του τι συμβαίνει στο Τιντούφ γνωρίζετε ένα στρατόπεδο προσφύγων στον κόσμο, έστω και ένα, όπου να μην έχει υπάρξει απογραφή, να μην έχουν ταυτοποιηθεί τα πρόσωπα, να αρνούνται ε, στην υπηρεσία ε, προσφύγων ε, του Ερυθρού Σταυρού, να δει ποιοι είναι οι πρόσφυγες αυτοί, γιατί είναι εκεί, πώς λέγονται, τι θέλουν να κάνουν. Τους το απαγορεύουν όμως. Όλα αυτά τα αποσιωπά φυσικά το συνενετικό κατά τα άλλα ψήφισμά σας. Εκνευρίζει η αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν να ακούν για καταστάσεις οι οποίες δεν είναι σωστές σε αυτά τα στρατόπεδα του Τιντούφ. Ποιος εφαρμόζεται στη χώρα, νόμος εφαρμόζεται στις, στους καταβλισμούς αυτούς. Ο νόμος της Αλγερίας ή ο νόμος του Πολυσάριο γιατί εμένετε τόσο πολύ ε, στο θέμα του δημοψηφίσματος. Και όταν κάποιος ε, αμφισβητεί το πρόσωπο, το, την ιδέα αυτή της ενιαίας της μοναδικής σκέψης, βλέπετε τι παθαίνει ο Σαλέ, δύο μήνες κράτηση και απέλαση μετά. Είμαι ειλικρινής μαζί σας, ε, είμαι παθιασμένος, αλλά αυτή είναι η άποψή μας για το συνενετικό σας ψήφισμα. Ήταν ένα βιαστικό ψήφισμα, Δικαιωμά σα βέβαια, εσείς πήρατε την απόφαση αυτή και κυρίως ε, ήταν άδικο απέναντι και στους νεκρούς, ήταν ένα άνισο ψήφισμα σε σχέση με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σας παρουσίασα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ δεν θα μπορέσω να δώσω το λόγο σε όλους τους συναδέλφους που το έχουν ζητήσει. Έχουμε ξεφύγει. Θα διαλέξω τρεις μόνο ανάμεσα στους εννέα είναι αφαίρετη η επιλογή μου, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο δίκαιος μπορώ. Γιάννε, σε ένα λεπτό. Ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, είναι αδύνατο μέσα σε ένα λεπτό να ασχοληθούμε με αυτό το τόσο περίπλοκο θέμα. Κύριε Υπουργέ, τρία ζητήματα. Καταρχήν σας ευχαριστώ που ήρθατε για τις ε, διευκρινήσεις που μας δώσατε. Αλλά ως προς την απεικιοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από, από Ή ε, κρεμεί και το θέμα της αυτοδιάθεσης με βάση τον ΟΗΕ. Τρίτον, η παγκόσμια κοινότητα και τα Ηνωμένα Έθνη είναι υπέρ του διαλόγου των εμπλεκομένων μερών. Βέβαια, μέσα αυτά τα 35 χρόνια, κάποια στιγμή είχατε δεχτεί την ιδέα του δημοψηφίσματος. Αλλά κάπου τελικά αλλάξατε γνώμη. Υπήρξε μια μεταστροφή εκ μέρους του Μαράκου. Δεν προεξοφλείται η έκβαση του δημοψηφίσματος αν θα είναι αυτονομία, αυτοδιάθεση, ανεξαρτησία ή τίποτε άλλο. Είναι πολύ δύσκολο κύριε Πρόεδρε μέσα σε ένα μόνο λεπτό. Και έχω και μια τελική παρατήρηση. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι αντιμαροκινικό. δεν ε, Μπορεί να έχουμε μεμονωμένους ευρωβουλευτές που να αντιδρούν κάπως εχθρικά απέναντι στο Μαρόκο, αλλά δεν διαπνέεται από τέτοιο πνεύμα κατά του Μαρόκου το συνενετικό ψήφισμα ίσως υπήρξε ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Νομίζω όμως ότι αυτό το πρόβλημα το καλύψαμε τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Δυστυχώς δεν μου επιτρέπει ο πρόεδρος να συνεχίσω. Διακόπτη ο πρόεδρος, ο κύριος Κασουλίδης, ένα λεπτό. Αφήστε με να ολοκληρώσω κύριε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, η Ισπανία δεν είναι δύναμη διοίκηση, δεν είναι διοικητική δύναμη με βάση το διεθνές δίκαιο και τα Ηνωμένα Έθνη. Κύριε Κασουλίδης, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω την παρουσία του Υπουργού και να πω τα εξή. Και στην επικράτεια της Δυτικής Σαχάρα και στα, στους του στρατού δεν υπάρχει επιτήρηση από τρίτους. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις ε, αποκλίνουσες απόψεις για τα γεγονότα. Λοιπόν, θα μπορούσε η κυβέρνηση του Μαρόκου να χρησιμοποιήσει τα δικά της ε, κυρίαρχα δικαιώματα να ορίσει μια επιτροπή από τρίτα μέλη που να μπορεί να πάει εκεί στη Δυτική Σαχάρα. Γιατί αλλιώς ο καθένας κάνει τα δικά του. Εμείς συζητήσαμε πολλές φορές εδώ το θέμα και βέβαια υπάρχει ε, πρόβλημα ότι ίσως οι πληροφορίες μας συλλέγονται με μη νόμιμους τρόπους, αφιβούλους τρόπους. Μπορείτε λοιπόν να ορίσετε ως κυβέρνηση του Μαρόκου μία επιτροπή από ανεξάρτητους εκπροσώπους που μπορούν να πάνε επί τόπου και να δουν ποια είναι η αλήθεια από όλες αυτές τις ιστορίες και τις εκδοχές που ακούγονται. Πρόεδρος, για να ολοκληρήσει η συζήτηση, ο κύριος ε, Παντσέρη, πρόεδρος της Επιτροπής Μαγκρέμ. Ένα λεπτό. Discusso con col fronte del Polisario sul senso della, della risoluzione. Σχετικά με τα σχόλια που έγιναν για το ψήφισμα. Κοιτάξτε, εμείς κάναμε μια προσπάθεια σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσουμε την διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία έχει ξεκινήσει στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Από την άποψη αυτή υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να υπάρξει αμέσως ένα ψήφισμα και σε άλλους που ήθελαν να περιμένουμε 15 μέρες. Εν πάση περιπτώσει τα πράγματα εξελίχθησαν όπως εσείς τα περιγράφετε κύριε Υπουργέ και νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα να επαληθεύσουμε επιτόπου μέσω μιας αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την κατάσταση. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε ανοιχτό τον διάλογο με το Μαρόκο γιατί είναι φυσικά σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει πρωταγωνιστικά στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ήδη τις ε, μικτές κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, ε, ίσως να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο, να δοθεί μια σαφής εντολή από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπάρξει επιτόπου έλεγχος της κατάστασης των πραγμάτων, από πλευράς μας υπάρχει η διαθεσιμότητα πλήρης. Κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε το λόγο για να κλείσετε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, δράση του Πρόεδρου Παντζέρη που έχει σημαντικό έργο με τους συναδέλφους ε, από, το, ε, τη Βουλή του Μαρόκο. σας ταυτόχρονα θα ήθελα να πω αυτό το σύστημα, αυτή η μεικτή επιτροπή δεν συνεδρίασει πριν να ε, υιοθετήσετε εσείς αυτό το ψήφισμα. Ίσως θα ήταν δυνατό να ακούσετε ή με τους δε να μοιραστείτε τις απόψεις αυτό το όργανο που είναι κεντρικό μέσω διαλόγου μεταξύ του Βουλή του Μαρόκου και του Ευρωβουλίου παρακολούθηκε. Λυπούμε γι' αυτό. Ταυτόχρονα εγώ πρότεινα να έρθω για μια ακρόση. Να προσπαθήσω να συμμεριστούμε τις απόψεις τους. Δεν ήταν δυνατό και αυτό. Με δική σας απόφαση. Είσαστε ανεξάρτητοι. Κυρίαρχοι να πάρετε ό,τι απόφαση θέλετε και να ψηφίσετε όποιο ψήφισμα. Αλλά χωρίς να ενημερωθείτε πριν. Δεύτερον, βέβαια η Ισπανία δεν είναι η διοικητική αρχή. Εδώ και μερικούς μήνες, εβδομάδες μάλλον θα έλεγα, τι βλέπουμε. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Ισπανία σαν διοικητική αρχή παίζει λίγο πάνω σε αυτό για την, ε, το θέαμα του Μαρόκου κλπ. Μα υπεγράφει διεθνή συμφωνία με την Ισπανία που κατατέθηκε. Παράνομα λέτε έτσι πιστεύετε. Εμείς όμως έχουμε διαπραγμάτευση με μια χώρα. Μια χώρα, ένα κράτος που υπέγραψε μαζί μας μια συμφωνία. Εσείς αποφασίσατε ήδη. Δεν θέλω να σας πείσω. Εσείς επαναλαμβάνετε τυφλά αυτά που λέει η Αλγερία και το Πολυσάριο. Δεν λέτε τίποτα για αυτούς. Εσείς βρήκατε τη λύση μαζί σας. Δεν πρόκειται να βρεθεί η λύση. Το Μαρόκο απα... Ε, ε, απαραίτητα θα βρίσκεται μέσα στο κέντρο μιας λύσης. Εσείς τώρα τι κάνετε, προσπαθείτε να δείξετε τον ουρανό. Αλλά ορισμένοι όταν σας δείχνουν τον ουρανό δεν κοιτάνε τον ουρανό, κοιτά το δάχτυλο που δείχνει τον ουρανό. Ε, μετά λέμε ε, γενοκτονία και λοιπά, α συγγνώμη, α, λάθος κάλαμε ε, χειρισμό από, το, από τους δημοσιογράφους. Α, όχι, λάθος. Μα κοιτάξτε, το σημαντικότερο είναι η διαπραγμάτευση. Μας προσφέρει θέλουμε να διαπραγματευτούμε και το κάνουμε. Αυτό ήθελα να σας πω. Όταν λέει ο όμως ότι εγώ εκπροσωπώ τον λαό των Σαραουή, εγώ λέω όχι, γιατί οι Σαραούι αλλιώς θα σκέφτονται, αλλιώς θα ζουν τα πράγματα η όρια αυτή ότι η λύση δεν μπορεί να βρεθεί παρά μέσω ενός δημοψηφίσματος. Μα προσπαθήσαμε να υπάρξει το δημοψήφισμα. Και αυτοί που λένε ότι μπορεί να βρεθεί το εκλογικό σώμα για να ε, ληφθεί μια απόφαση ψεύδονται. Ψεύδονται. Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε. Διαπραγμάτευση. Υπενθύμησα τους όρους του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με ακρίβεια. Η αυτοδιάθεση θα πρέπει να βρεθεί μέσω διαπραγμάτευσης και της αναζήτησης μίας πολιτικής λύσης. Ας λαωθούν υπόψη οι σοβαρές προσπάθειες που κατέβαλε το Μαρόκο βάσει συμβασμού, βάσει ελελεσμού. Εμείς με αυτή την καλή πίστη μπήκαμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις. Μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων όμω, όταν ο ειδικό απεστασμένο των ε, Ηνωμένων Αθηνών είπε ότι η επιλογή τη ανεξαρτησία δεν είναι αναλυστική, τα πετάξαμε έξω. Μετά που έκανε τέσσερι γύρου στην ε, στην περιοχή που προέδρευσε τεσσάρων συνεδριάσεων διαπραγμάτευση. Πήραν άλλον και αρχισαν πάλι από το μηδέ. Προσπαθώντα στην Όρκη να αλλάξει η μέθοδο διαπραγματεύσεων, να επιταχθεί ο ρυθμό και να περάσουν σε καινούριε διαδικασίε. Ελπίζω όμω αυτέ οι νέε διαδικασίε διαπραγμάτευση θα μα επιτρέψουν να επιταχύνουμε πραγματικά το ρυθμό. Γιατί ο στόχο δεν είναι το δάχτυλο που είπαμε που δείχνει, είναι ο ουρανός. Ο στόχος είναι μια συμφωνία στην οποία θα συμφωνήσουν όλοι. Λοιπόν, γιατί να υπάρχουν όροι εάν βρούμε μια συμφωνία βάση της διαπραγμάτευσης. <clears throat> Κανένα δεν διαπραγματεύεται όταν οι διαπραγμάτευτε γίνονται υπό τον όρο ότι οπωσδήποτε πρώτα θα πρέπει να υπάρξει το δημοψήφισμα. Όπω γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλγερία. Λυπούμε πως είναι συνάδελφος μου Αλγερινός δεν είναι παρόν. Λυπούμε γιατί είναι διάλογος. Όπως έχουμε και μαζί σας. Πρέπει να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα, ανοιχτά, ειλικρινά. Λυπούμε που δεν είναι εδώ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να υπάρχει το Μακρέπ να μας βοηθήσει η Αλγερία να βρούμε μια λύση. Να μας βοηθήσει, λέω, η Αλγερία να βρούμε λύση. Γιατί θα προτιμούσα να είναι παρόν λόγω του ότι η Αλγερία είχε εμπλεκεί Πολέμησε με το στρατό της Αλγερίας στις ε, περιοχές αυτές, το ξεχάτε. Πήρε ε, ε κρατούμενος από τον Μαροκινό στρατό. Το ξεχνάμε αυτό. Η Αλγερία είναι υπεύθυνη για αυτό που γίνεται στη δική της επικράτεια και ιδίως μέσα στα πλαίσια της συνθήκης της Γενέβης, της ευθύνης το, για να υπάρχουν οι πρόσφυγες εκεί στο εδάφι Δεν έχουν δικαίωμα να πάνε οι άνθρωποι αυτοί να εργαστούν σε όλη την επικράτεια της Αλγερίας. Δεν θεωρούνται άτομα. Γιατί, γιατί, γιατί. Να το συστήσουμε όλα αυτά με τον Υπουργό της Αλγερίας. Καμιά φορά το κάνουμε στα παρασκήνια κάποια συνάντηση. Το κάνουμε καμιά φορά και μέσα στα πλαίσια των ΗΠΑ λόγω της ευθύνη που φέρει η Αλγερία. Και τέλος, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτό που ξέρουν μεταξύ ημών <clears throat> ότι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος πληρώνει για την ε, υποστήριξη των προσφυγικών πληθυσμών αυτών. Επενδύεται εκεί. Να επενδύσετε κάτι παραπάνω σε αυτά που κάνει η Κομισιόν όμως και στα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η Κομισιόν όσον αφορά την επιστική βοήθεια που δίνει. Η μόνη αναφορά στους πρόσφυγες που έχετε στο ψήφισμά σας είναι η ε, ανθρωπιστική βοήθεια, χωρίς να βοηθήσετε στο νομικό καθεστώς, στο, στο δικαίωμα να υπάρχουν επί χάρτου στο δικαίωμα της ε, <clears throat> επιστροφής ε. αν οι άνθρωποι αυτοί να να ζούσουν αλλού. Τι κάνετε εσείς, ποιος σας λέει ότι όλοι μένουν εκεί γιατί έχουν μία έμονη ιδέα, την ίδια. Γι' αυτό παραμένει σίγουρο το Μαρόκο ότι μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων, γιατί θέλει να βρει τη λύση, θα μπορεί να βρεθεί η λύση εκεί. Και γι' αυτό δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα της ε, διάσπασης. Να μην εγκαταλείψουμε τις βασικές ιδέες. Θα πρέπει να έχουμε κάποιες δράσεις που γίνονται, δίκαια κλπ, να τις αντιμετωπίσουμε έναντι μιας προπαγάνδας η οποία εκμεταλλεύεται κάποιες δυνάμεις ιδίως στην Ισπανική. Γνωρίζετε το Reuters, την Washington Time και άλλες σοβαρές εφημερίδες που πήγαν εκεί. Πήγαν εκεί επί τόπου και το και να φύγουν. Γιατί δεν ήρθανε μέσω μιας αποκριστικής ισπανικής πηγής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παραμένουμε σε επαφή, ελπίζουμε η Μικτή Επιτροπή να συνεδριάσει πολύ γρήγορα. Η κυβέρνηση πρόφανως παραμένει στη διάθεση της Επιτροπής Εκτορικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυόμιση εκατομμύρια Μαροκανοί εξέφρασαν αυτή την, ε, την βούληση μετά από μία πρόσκληση σε μία πορεία 48 ωρών στην Καζαμπλάνκα. Αυτή είναι η αντίδραση της κοινή γνώμη στο Μαρόκο, συμπεριλαμβανομένου και των συνολών που έλαβαν μέρο στην πορεία αυτή. Σήμερα μας ζητάτε τους λογαριασμούς ότι γιατί χρησιμοποιήσετε ένα ε, Χρησιμοποιήστε ρόπαλο, τα ξέρετε ότι υπήρχαν από την άλλη μεριά μαχαίρια, βόμβες μολότοφ κλπ. Σήμερα μας κατηγορούν εμά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ζητώ συγγνώμη για μια ακόμη φορά από συναδέλφου που δεν μπόρεσαν να πάρουν το λόγο. Ο διάλογος θα συνεχιστεί σε μια δύσκολη ε, κατάσταση και σε μια περίπτωση ευαίσθητη. Θα υπάρξει ελπίζω μια άλλη συνάντηση σε ένα λιγότερο πολεμικό και ευαίσθητο κλίμα και χωρίς ανθρώπινα θύματα. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Υπουργό, ένα λεπτό διάλειμμα και περνάμε στο επόμενο θέμα. E Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και γι' αυτό χωρίς πολλά εισαγωγικά μπορούμε νομίζω να ξεκινήσουμε την εξέταση της πρότασης ψηφίσματος για την Κροατία. Λυπάμαι, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Σβόμποντα, ο οποίος δέχτηκε να καθυστερήσει η συζήτηση για το ψήφισμά του, αλλά α, θα ξεκινήσει με πάρα πολλούς θορύβους, τους οποίους δεν μπορώ εγώ να μειώσω. Θέλω να ζητήσω μόνο από όλους εσάς να φύγετε εκτός εθούσης. Κύριε Σβόμποντα, έχετε το λόγο. Ah, ah, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνω, λοιπόν, ότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα υπάρχει αναβολή. Ε, ευτυχώς δεν είναι τόσο αφιλεγόμενη η Κροατία όσο και η... το θέμα της Σαχάρας. Ε, γι' αυτό θα είμαι και σύντομος. Θα αναφερθώ στα πιο σημαντικά σημεία. Καταρχήν, θα ήθελα να τονίσω ότι η Κροατία, ιδίως στους τελευταίους μήνες, κατέβαλε σημαντικότητε προσπάθειες για την επιβολή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Δεν ήταν πάντα εύκολα τα πράγματα και ορισμένοι από του επιτρόπου πολιτικούς επίσης δυσκολεύουν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, η κροατική κυβέρνηση έχει θέσει σωστού όρου όσον αφορά κυρίω η δικαιοσύνη και την καταπολέμηση διαφθορά. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Γιατί αν δω και τη χώρα μου την Αυστρία βλέπω ότι υπάρχει εύρια συνένεση για την ένταξη τη Κροατία. Υπάρχουν όμως και ανησυχίε όσον αφορά το θέμα της καταπολέμησης της ε, διαφθοράς. Ε, στην Κροατία θα εξεταχθεί το Μάρτιο αν έχει φτάσει στα benchmarks και ελπίζω ότι θα είναι ανοιχτή για τον έλεγχο αυτό η Κροατία. Ένα πρόβλημα είναι η συνεργασία με το Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη. Ελπίζω ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια η Κροατία ούτως ώστε να βελτιστοποιήσει, να μεγιστοποιήσει θα έλεγα μάλιστα αυτή τη συνεργασία. Τι το θέμα κατά πόσον υπήρξαν τα έγγραφα αυτά, κατά πόσον καταστράφηκαν. Ε, θα πρέπει να επιληθεί το θέμα γιατί δεν υπάρχει υπόλοιτη έλλειψη συνεργασίας, ίσως υπάρχει κάποιο μικρό κενό, αλλά ελπίζω ότι θα υπάρχει συμφωνία των Υπουργών Δικαιοσύνης για την ολοκληρώση αυτής της συνεργασίας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα και ε, εμπόδιο για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, τι το θέμα του ανταγωνισμού σε σχέση με τα ναυπηγεία. Θα πρέπει να πούμε ότι σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση δεν φτάνουμε στην βέλτιστη λύση. Η κροατική κυβέρνηση γνωρίζει, νομίζω ότι αυτά χρειάζονται. Πρέπει από την άλλη μεριά να φροντίσουμε η μεταρρύθμιση των ναυπηγείων να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην οδηγεί σε νέα προβλήματα. Τις περιοχές εκεί. Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι η συνεργασία μεταξύ Ελφίας και Κροατίας βελτιώθηκε σημαντικότατα αναφέρεται αυτό. Οι δύο πρόεδροι ανέλαβε σημαντικέ προσπάθειε και χαίρομαι που ο πρόεδρο Στάβιτ ήταν ακριβώ στη Βουκοβά τελευταία και αναγνώρισε τα εγκλήματα που έγιναν εκεί. Ήταν σημαντική πληγή αυτή που προς την Κροατία. Είχα πάει μετά αμέσως την ένταξη αυτή με την ε, Doris Pack υπάρχουν έτσι σημαντικά, γίνονται σημαντικά πολιτικά βήματα παραδείγματος χάνει δημιουργία ενός μνημείου. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ για το θέμα των μειονοτήτων. Καμία χώρα δεν έχει λύσει πλήρως το θέμα των μειονοτήτων. Η εντύπωση μου είναι ότι το θέμα των μειονοτήτων ε, προχωράει, ε, υπάρχουν πολλές προσπάθειες που καταβάλλονται. Βέβαια η ενσωμάτωσή τους δεν είναι δυνατή, εύκολη θέλω να πω σε αυτές τις, ε, τους καιρούς της κρίσης, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να καταβληθούν πάρες πολλές προσπάθειες όσον αφορά το θέμα της στέγασης, ιδίως της κοινωνικής στέγης, προβλήματα υπάρχουν ακόμα που είναι προβλήματα που μπορούν να επιληθούν. Τελευταία παρατήρηση, πώς θα προχωρήσουμε. Είμαι σε στενή συνεργασία με την Ουγγρική Προεδρία και με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρτων, με τον οποίο συνομίλησα πρόσφατα. Έχουμε κάθε συμφέρον η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας, δηλαδή το πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτους. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να εγκρίνει το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας, ίσως στη Σύνοδο του Ιουλίου το επόμενο έτους θα είναι και αυτό πολύ δύσκολο. Παρ' αυτά θα προσπαθήσουμε η διαδικασία στο Κοινοβούλιο χωρίς να αμελήσουμε κάτι <laughs> να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο τόσο ώστε να μπορούμε έγκαιρα να αρχίσουμε διαδικασία επικύρωσης ούτως ώστε ιδανικά να γίνει η ένταξη την 1η Ιανουαρίου 2013 ή τουλάχιστον κατά διάρκεια του 2013 για να μπορέσει να ωφεληθεί η Κροατία και να συμμετάσχουν οι Κροάτες στις ευρω... Ε, εκλογές του 2013. Αλλά γίνονται πολλά από τις κυβερνήσεις και στη Σλοβενία, Σλοβενία συγγνώμη, και στην Κροατία, ούτως ώστε στη Σλοβενία να υπάρχει ένα θετικό κλίμα τώρα για τη γειτονική χώρα Πολλά πρέπει να κάνουμε και είμαι πεπισμένος ότι αυτά θα γίνουν σωστά και πλήρως και γλίγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σπόσελτ, δύο λεπτά. Ja, Herr Präsident, also ich kann dem äh, mündlichen Vortrag des Kollegen ε, πρόεδρε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την προφορική παρουσίαση του κυρίου Σφόβοτα. Ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε γενικέ γραμμέ με το κείμενο που έχουμε μπροστά, παρόλο που πρέπει να δούμε τι γίνεται σε ορισμένα σημεία, ιδίω στη διατύπωση στα σημεία 6 και 11, στα οποία αναφέρθηκε και ο κύριο ε, ε, Σφόμποτα, δηλαδή ε, διαφθορά και συνεργασία με την ΕΚΤΗ. Πραγματικά θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία, να ασκήσουμε κριτική εκεί που είναι δικαιολογημένη. Απ' την άλλη μεριά όμως να πούμε ξεκάθαρα ότι υπήρχε σημαντική πρόοδος και ότι πραγματικά προσπαθεί η κυβέρνηση να προχωρήσει στους προβληματικούς τομείς. Και αυτό είναι νομίζω καλή παιδαγωγική να αναφερόμαστε δηλαδή και στις θετικές εξελίξεις. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του κυρίου Σφόμποντα, θα ήθελα να αναφερθώ σε λίγες από αυτές. Καταρχήν, Ουγγρική Προεδρία. Έχουμε δηλώσει και από την Κομισιόν και από την Ουγγρική Προεδρία ότι θέλουν οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Στο Κοινοβούλιο εμείς θα πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη και να τα υποστηρίξουμε. Να τονίσουμε δηλαδή ότι και τα δύο αυτά όργανα έχουν αυτό το στόχο. Ταυτόχρονα νομίζω ότι η συνένεσή μας θα πρέπει κατά δυνατόν να δοθεί τον Ιούλιο η σύμφωνη γνώμη μας θα ήταν έτσι ένα σημαντικό μήνυμα στην διαδικασία επικύρωσης στα κράτη-μέλη, ότι εμείς δρούμε χωρίς καθυστέρηση και ότι καλούμε και τους άλλους να δράσουν επίσης χωρίς καθυστέρηση. Όσον αφορά τη διαδικασία επικύρωσης, διαπραγματεύσει δηλαδή να ολοκληρωθούν στο πρώτο εξάμενο, κατά δυνατόν τον Ιούλιο να επικυρώσουμε εμεί και μετά θα αρχίσει η διαδικασία επικύρωση. Και όσον αφορά αυτή τη διαδικασία, θα ήθελα να σα πω ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να φροντίσουμε οπωσδήποτε να μην εμπλακούν ξένα στοιχεία στη διαδικασία αυτή τη επικύρωση που θα μπλοκάρουν τη διαδικασία. Ίσως ξένα στοιχεία που θα επιταχύνουν τη διαδικασία σε αυτό, αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν προσεκτικά. Το να πούμε ναι δεν θα ολοκληρώσει τη διαδικασία είναι σημαντικό να μπορέσουμε να επιδράσουμε θετικά και στη διαδικασία επιχείρηση. Δυστυχώ δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Τελειώνω, Πρόεδρε. Θα ήθελα όμω να πω ξεκάθαρα ακριβώ όσον αφορά τα λεπτά θέματα, δηλαδή η συνεργασία στον τομέα τη δικαιοσύνη, καταπολέμηση της διαφθοράς και έκτης, η Κροατία τους τελευταίους μήνες προχώρησε σημαντικότατα και θα πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα. Νορεβόλε Βάιγκολ δύο minuti. Spoštovani gospod predsedujoči. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σβόβοντα, όπως πάντα, συνέταξε μια ρεαλιστική και καλοπροαίρετη έκθεση που μπορεί να υποστηριχθεί από την ομάδα σχεδόν σε όλα τα σημεία. Υπάρχουν κάποιες μικρολεπτομέρειες που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε, αλλά με το σύνολο της έκθεσης συμφωνούμε. Είναι πολύ καλή και ισορροπημένη και ευελπιστούμε ότι η, Κροατία θα γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη στιγμή που θα συμμορφωθεί με όλα τα κριτήρια. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμη και η κροατική κυβέρνηση αλλά και το, ο λαός της Κροατίας θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν. Δεν είναι όλοι οι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, οι λεωφόροι. Μερικές φορές το οδόστρωμα έχει τρύπες και θα πρέπει να τις διορθώσουμε. Στην κρατή αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα κλίμα που χαρακτηρίζεται από την ε, οικονομική κρίση και έχει προκαλέσει μία αποκαρδίωση του κρατικού λαού και μία αποδυνάμωση της προηγούμενης θερμής υποστήριξης που έδειχνε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πάντως που είναι σημαντικό είναι ότι υπήρξε μια πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα στο θέμα των σχέσεων γειτονία. Ε, η Κροατία εγγενίασε ένα νέο πολύ ευίωνο κεφάλαιο στη σχέση της με τη Σερβία και ο πρόεδρος Τάντιτς δεν επισκέφθηκε μόνο το Βούκοβαρ για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα του απολυταρχικού καθεστώτος του Μιλόσεβιτς, αυτό που ήταν ακόμη πιο σημαντικό κατά τη γνώμη ήταν όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι, ο Κροάτης πρόεδρος Ιωσίποβιτς, εξέφρασε και αυτό στη θλίψη του για τα σερβικά θύματα αυτής της ένοπλης σύραξης. Σε ό,τι αφορά τα μέσα, την ελευθερία έκφρασης, το μέσο μαζικής ενημέρωσης, την ελευθεροτυπία και τους δημοσιογράφους. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το προσέξουμε. Το ίδιο ισχύει και για τις μειονότητες, για τους ομοφιλοφίλους, αλλά και για άλλες μειονότητες. Δεν μιλώ μόνο για αθηνοτικές μειονότητες. Οι μειονότητες γενικώ είναι ένα κρεμές θέμα στη σχέση με την Κροατία. χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Θα ήθελα <coughs> να συγχαρώ τον κύριο Σφόμποντα για το πολύ αξιόλογο ψήφισμα και να εκφράσω την αμύωτη υποστήριξή μας ε, στην ενταξιακή προοπτική και διαπραγμάτευση της Κροατίας. Και ελπίζω η κόποση της διεύρυνσης να μην υπονομεύσει την υποστήριξη του κρατικού λαού. Φυσικά θα πρέπει η Κροατία να εκπληρώσει όλα τα κριτήρια και τα τους συγκριτικούς κανόνες και ελπίζω να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα της ένταξης. Όπως είπατε, μέχρι στιγμής εφαρμόστηκαν πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Το επισήμανε και ο κύριος ε, Σφόβοντα. Είχαμε πρόοδο και στην περιφερειακή συνεργασία. Αναφερθήκατε στην πρόσφατη επίσκεψη του, Προέδρου, του Σέρβου Πρόεδρου Τάντιτς στο Βούκοβαρ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Επίσης, ε, υπάρχουν ε, σημαντικοί τομείς όπως η πράσινη ενέργεια και οι δημόσιες συγκοινωνίες που είναι τομείς ε, ιδιαίτερα πρόσφοροι για διαπεριφερειακή συνεργασία. Βέβαια, διαπιστώνουμε και κάποιες αδυναμίες και κάποιες ελλείψεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα σημαντικό θέμα είναι η αμεροληψία της δημόσια <coughs> διοίκησης. Θα πρέπει αυτό το θέμα να ενισχυθεί, να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης Κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολική η συνεργασία της δικαιοσύνη με το κυβερνόν κόμμα και φυσικά να αναβαθμιστεί και ο αγώνας για την πάταξη της διαφθοράς και το θέμα της χωροταξίας, ε, πολεοδομίας και διαχείρισης των πόρων ε, θα πρέπει να προσεχθούν. Πολύ σημαντική τομή. Αναφέρθηκε το θέμα της ε, καταπολέμησης των διακρίσεων. Είναι σε καλό δρόμο, αλλά θα πρέπει να ενταθεί αυτός ο αγώνας. Όντως διαπιστώσαμε μία αποδυνάμωση της ε, υποστήριξης ε, του λαού για την ένταξη της Κροατίας. Ήταν σωστή αυτή η επισήμανση. Αυτό δεν οφείλεται μόνο σε, στην πολιτική της κυβέρνησης ε, του Ζάγκρεπ. Είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσπαθεί να αναμίξει πιο ενεργά την κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για πιο ενεργό ανάμειξη των ε, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και εν ώψη και του δημοψηφίσματος θα πρέπει να ε, εντατικοποιήσουμε μια διαδικασία δημοσίων σχέσεων. Κύριε Κοπά, για δύο λεπτά. Θέλω να εκφράσω συγχαρητήρια στον συνάδελφο Σβόμποντα για την απόλυτα ισορροπημένη έκθεση που επιβεβαιώνει την επιθυμία του Κοινοβουλίου γιατί όσο το δυνατόν γρηγορότερη ένταξη της Κροατίας στην Ένωση και παράλληλα δείχνει τα εναπομείναντα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Είναι πράγματι σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτή την προσέγγιση, εκφράζοντας την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μπήκαν πια στο τελικό του στάδιο. Ε, ένα σημείο θέλω να αναφέρω, το οποίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό και αφορά τη διαδικασία συμφιλίωσης και ειδικότερα το ζήτημα της επιστροφής των προσφύγων του πολέμου στην Κροατία, ζήτημα σημαντικό που υπάρχει στην έκθεση. Ε, θέλω να αναφερθώ στη συμφωνία η οποία έγινε πρόσφατα ανάμεσα στους προέδρους της Σερβίας και την, της Κροατίας για την αποκοινού αντιμετώπιση του ζητήματος των προσφύγων και ε, από την οποία συνάντηση ακολούθησαν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Έχει πράγματι σημασία να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες και να τονίσουμε ότι η Κροατία πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες για την επιστροφή των Σέρβων υπηκών τη, μια επιστροφή που θα πρέπει να φροντίζουμε να υποστηρίζεται από μέτρα που θα εγγυώνται τη βιωσιμότητα ε, αυτής της διαδικασίας των ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν. Ε, θέλω να τελειώσω με μια ευχή να είναι η τελευταία έκθεση πρόοδου για την Κροατία που επεξεργαζόμαστε και σύντομα να έχουμε τους Κροάτες συναδέλφους στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κοπά. Ο κύριος Στάνο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια κύριε Σφόμποντα εκ μέρου τη ομάδα μεταρρυθμιστών και συντηρητικών και εμεί είμαστε υπέρ τη διεύρυνση προ τα Δυτικά Βαλκάνια και φυσικά η Κροατία είναι σε πολύ προηγμένο στάδιο προενταξιακό. Όπω ανέφεραν και προλαλήσαντε, υπάρχει συνένεση στην Επιτροπή μα ότι θα πρέπει στην Κροατία και το κράτος δικαίου και η πάταξη της διαφθοράς, ακόμη και στα υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης, να τεθούν ως ύψιστη προτεραιότητα. Σε προηγούμενες διαφερήνσεις δεν είχε αντιμετωπιστεί δεόντως αυτό το θέμα, να μην επαναλάβουμε το ίδιο σφάλμα, ε, αν θέλουμε να πείσουμε το ευρωπαϊκό κοινό ότι η διεύρυνση είναι θετικό. Χαίρομαι για την επίσκεψη του Σέρβου Πρόεδρου στο Βούκοβαρ και για, το, για την ε, επίλυση της συνοριακής ε, διαμάχης με τη Σλοβενία, γιατί ήταν ένα θέμα που επισκίαζε την ενταξιακή διαδικασία. Ελπίζω να ασχοληθεί και με το θέμα των μειονοτήτων η Κροατία, ιδιαίτερα της σερβικής μειονότητα. Σίγουρα η Κροατία θα είναι η επόμενη χώρα που θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός και αν γίνει κανένα θαύμα και την προλάβει η Ισλανδία. Πάντως η Κροατία και η είναι αυτή τη στιγμή οι μόνες υποψήφιες χώρες που κατά πάσα πιθανότητα θα ενταχθούν μέσα στο επόμενο 18 μήνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει πάντως εμεί ως πολιτικοί να εξηγήσουμε τις θετικέ πτυχές αυτή τη ε, διεύρυνση στους ψηφοφόρους μα. Στην πατρίδα μου ε, υπήρξε μια μεγάλη και ξαφνική εισρωή μεταναστών που δημιούργησε πολλές ε, ταραχές και φοβερό σκεπτικισμό, ιδιαίτερα των ε, ε, κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της διεύρυνσης. Θα πρέπει λοιπόν να προσετεριστούμε τους πολίτες ότι δεν θα υπάρξουν απειλές όπως αυτές που δημιουργήθηκαν στην αγορά απασχόληση του Ηνωμένου Βασίλειου για να συμφωνήσει και το κοινό με τη διεύρυνση. Ο κύριος Ντανζόν, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ θερμότατα τον κύριο Σβόμποντα για την ε, εξαιρετική του έκθεση. Και μάλιστα, ενώ μερικέ φορέ οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων αμφιβάλλουν για το κατά πόσο είναι εφικτό, αφικτή αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική που τους προσφέρουμε εδώ και μια δεκαετία, καλό ήταν να επιμένουμε και στις θετικές πτυχές και στις ε, επιτυχίες ορισμένων χωρών όπως της Κροατίας που είναι σε πολύ καλό δρόμο και ελπίζω να ενταχθεί το συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα για όλη την περιοχή και έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα και είναι ενθαρρυντικό και για τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Όπως είπαν ε, και οι συνάδελφοι είναι πολύ ενθαρρυντικά αυτό που συμβαίνει με, στην βελτίωση των σχέσεων με την Σερβία. Και πέραν των εικόνων που και αυτές είναι πολύ σημαντικές για την παρουσία του Πρόεδρου Τάντιτ στο Βούκοβαρ, Πίσω από αυτές τις επαφές όμως και συνομιλίες κρύβονται πολύ σημαντικές πρόοδοι που έγιναν για ευαίσθητος τομείς, αγνοούμενους, πρόσφυγες, δικαιώματα κυριότητας, ανάκτηση περιουσιών κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και αυτή η ενέργεια που δείχνουν οι πολιτικοί Ιωσίποβιτς και Τάντιτς είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να έχει αντίκρισμα, έχει αντίκρισμα και στην κοινωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αποθάρρυνση ή την ψυχρότητα που αρχίζει να δείχνει ο κρατικός λαός απέναντι στη διεύρυνση, ελπίζω ότι δεν είναι επανόρθωτη αυτή η απώλεια του ενθουσιασμού και ελπίζω να αντιστρέψουμε αυτή την ψυχροτητα που αρχιζει να δειχνει ο κρατικο λαος απεναντι στη διευρυνση ελπιζω οτι δεν ειναι επανορθωτη αυτη η απωλεια του ενθουσιασμου και ελπιζω να αντιστρεψουμε αυτη την ταση όπως είπε και η κυρία Βαρκαδέ, θα πρέπει να δούμε τι μηνύματα στέλνουμε προς την κοινωνία των πολιτών και προς την Κροατία γενικά. Γιατί μερικές φορές, κατά την έναρξη των διαπραγματευτικών κεφαλαίων, ήμασταν υπερβολικά δυσανάλογα απαιτητικοί απέναντι στην Κροατία και ανισόρροπα μερικές φορές. Και αυτό έδωσε πολύ κακή εντύπωση, πολύ κακή εντύπωση στον κρατικό λαό. Θα πρέπει λοιπόν με παιδαγωγικό τρόπο να τους ε, επαναφέρουμε την ουσιαστική και γνήσια ελπίδα της ε, προσχώρησης. Σας αποκάλεσα αντιπρόεδρο της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνα. Συγγνώμη, είστε πρόεδρος της Υποεπιτροπής και όχι αντιπρόεδρο. Ο κύριος Κάτσιν, για ένα λεπτό. Η Κροατία Κυρίε και κύριοι, ένα πολύ σημαντικό παίκτη ε, στην κατάσταση των Δυτικών Βαλκανίων. Και το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλούμε για την εξασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή και τις ε, αγαστές ε, σχέσεις μεταξύ γειτονικών χωρών. Ευχαριστούμε τον κύριο Σφόμποντα γιατί είναι πολύ ισορροπημένη η έκθεσή του πιστεύω ότι μπορούμε να εντείνουμε την υποστήριξή μας προς την Κροατία για να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις. Τον επόμενο Ιούνιο θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από τότε που η Κροατία και η Σλοβανία ε, Σλοβενία ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους. Ήταν μια πολύ σημαντική καμπή και για τις δύο χώρες. Και ένα εξάμεινο αργότερα θα συμπληρώσουμε 20 χρόνια από τη διεθνή τους αναγνώριση ως ανεξάρτητες χώρες. Στην Κροατία Υπάρχει συνένεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το θέμα αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την όθηση που έχει δημιουργηθεί για να διεκπαιρεώσουμε αυτή την ενταξιακή διαδικασία. Η έκθεση αναφέρεται στην ανάγκη οριοθέτηση των συνόρων. Διαφωνώ, Χάνες, με την διατύπωση αυτή. Γιατί όταν λέμε συνοριακή οριοθέτηση είναι ένα πολύ τεχνικό θέμα και στα Δυτικά Βαλκάνια τίποτα δεν ε, πραγματοποιείται χωρίς ε, πολιτική ε, βούληση και χωρίς βελτίωση του πολιτικού κλίματος. Έγινε μια συμφωνία διαιτησίας ως προς τα σύνορα, οπότε από τεχνική άποψη έχει βρεθεί λύση, αλλά χρειάζονται και πολιτικές προσπάθειες και αντίστοιχη πολιτική βούληση χρειάζεται και στις σχέσεις με τα υπόλοιπα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό. Τέλος, μία μικρή προειδοποίηση. Φαντάζομαι ότι όλοι οι Σλοβαίνοι ευρωβουλευτές θα εγκρίνουν την έκθεση Σφάμποντα. Πριν από μισό χρόνο υπήρξε, υπήρχε διχασμός, διάσταση μεταξύ μα. Μόνο οι μισοί ήμασταν υπέρ τη Έκθεση προόδου, ενώ οι άλλοι μισοί για πολιτικού λόγου ήταν κατά. Εγώ πιστεύω ότι τώρα υπάρχει πρόσφορο έδαφο και συνένεση μεταξύ των Σλοβαίνων Ευρωβουλευτών και θα υποστηρίξουμε όλη την έκθεση. Ο κύριο Πέτερ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαρώ τον συνάδελφο Σφόμποντα για την πολύ καλή έκθεση που και εγώ θα υπερψηφίσω και συγχαίρω και την Κροατία για την εντυπωσιακή πρόοδο που πραγματοποίησε στις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Κροατία έχει το δυναμικό να συνεχίσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και να κρατήσει ε, την ορμή που έχει και τον ενθουσιασμό και στην τελευταία φάση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η έκθεση αναφέρεται και στο συνοριακό ζήτημα. Άκουσα ένα προλαλήσαντα και θα ήθελα να πω ότι η Σλοβενία και η Κροατία δεν έχουν καταλήξει σε οριστική ε, λύση <clears throat> για το θέμα των συνόρων. Απλώς αποφάσισαν πώς θα προχωρήσουν στην οριστική λύση όταν δημιουργηθούν ε, οι προϋποθέσεις. Αλλά είναι, δεν υπάρχει ακόμη τέτοια οριστική λύση για το συνοριακό. Επίσης συμφωνώ με όσους είπαν ότι και οι δύο χώρες, ακόμη και με τη χρήση της ρήτρας της Συμφωνίας Διατησίας, μπορούν να ε, να χρησιμοποιήσουν ε, διμερείς προσπάθειες για να βελτιώσουν την αμοιβαία τους εμπιστοσύνη, γιατί εκεί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Και στη Σλοβενία υπήρχε διχασμός. Ο κυβερνητικός συνασπισμός κέρδισε το δημοψήφισμα, αλλά πολύ ωριακά. Δεν είμαστε λοιπόν βέβαιοι για την ε, οριστική λύση γιατί τι ακριβώς περιεχόμενο θα έχει. Οι κυβερνήσει βέβαια δεν θα πρέπει να στηρίζονται σε προτάσει ε, έξωθεν. Θα πρέπει να φροντίσουν με κοινέ προσπάθειε και αμοιβαία εμπιστοσύνη να καταλήξουν σε ένα συνενετικό κοινό αποτέλεσμα που θα τηρεί το, το ευρωπαϊκό πνεύμα και θα βελτιώνει τις διμερείς σχέσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πακ για δύο λεπτά. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο Σόβοντα Μπορώ απόλυτα να συμφωνήσω με τα περισσότερα σημεία της έκθεσής του. Μάθαμε όμως από την εμπειρία με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά το θέμα ακριβώς της διαφθοράς και είμαστε πιο αυστηροί έναντι της ε, Κροατίας και ίσως τα σημεία 6, 7 και 8 θα μπορούσαν να τροποποιηθούν ούτως ώστε να τονιστεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος πολύ περισσότερο από ότι οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Και επίσης θα ήθελα να πω, ορισμένοι συνάδελφοι είπαν ότι πριν από 20 χρόνια πήραν την ανεξαρτησία τους και δύο χώρες και η μία από τις δύο χώρες είναι ήδη μέλος από το 2004 και θα ήταν καλό εν ε, αυτή η χώρα προωθούσε την ένταξη Κροατίας με ενθουσιασμό. Υπάρχουν ε, περισσότερες αντιδράσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κροατία. Το ξέρω αυτό, είναι κάτι που γίνεται σε πολλές χώρες που οι διαπραγματεύσεις διαρκούν τόσο πολύ. Αυτά οφείλονται στη μακροχρόνια διαμάχη με την Σλοβενία και στην σχετικά άδικη στάση ε, του κυρίου κατηγορού όσον αφορά την ε, συνεργασία της Κροατίας με στα πλαίσια ΣΥΚΤΗ του Διεθνούς Ποινικού ε, Δικαστηρίου. Γιατί ε, συζήτηση για κάποια έγγραφα τα οποία εμείς δεν ξέρουμε καν σίγουρα όπως είπε και ο κύριος ε, υπάρχουν. Θα πρέπει απλώς να τους πούμε ότι είναι σωστή η οδός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε όχι με προπαγάνδα αλλά με φιλική στάση και όντας ε, φιλική προς εκείνους που εργάζονται σκληρά στη χώρα αυτή και λαμβάνουν αποφάσεις που ήταν πάρα πολύ δύσκολες για τους πολίτες. Ελπίζω λοιπόν από κοινού να πετύχουμε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το επόμενο έτος, μέσα του έτους, ούτω ώστε να μπορούμε ήδη από το φθινόπωρο του χρόνου να έχουμε Κροάτες παρατηρητές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Λίγο ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει ο κ. Χάουιτ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι ε, θα ρίνουμε εμείς τους κράτες ε, στην μελλοντική τους ε, ένταξη. Θα ήθελα να πω σεβόμαστε το δημοψήφιο στη Σλοβενία παρόλο που συμφωνώ ότι ελέγχθη ότι πολλά μπορούν να γίνουν. Παρόλο που έχει έρθει το εμπόδιο για την πρόοδο και συγχαρώ λοιπόν τους Σλοβένους. Θα ήθελα να συγχαρώ τον φίλο Σβόμποντα για το έγγραφό του και την έκθεση που υποβάλλει. Ε, βέβαια είναι σημαντικό αυτό που λέγεται για σεβασμό του ΙΚΤΗ. Και επίσης το θέμα ότι θα πρέπει να γίνεται ε, ε, ενδεχομένως να δικαστούν οι άνθρωποι αυτοί για εγκλήματα ε, πολέμου στις ίδιες τις χώρες. Ε, οι παράγραφοι 9 και 13 του κειμένου χαίρομαι που υπάρχει πρόοδος και πραγματικά ε, συμφωνώ με το κείμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Λάγκε θέλει να πει κάτι, δύο λεπτά. Δεν έχουμε πάρα πολύ περισσότερο χρόνο. Thank you very much, Chairman. Just to inform you that... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή μόλις προετοίμασε αρχές Νοεμβρίου μία έκθεση προόδου, στα πλαίσια της οποίας η Κομισιόν εκτιμά θετικά γενικά τις εξελίξεις στην Κροατία και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι διαπραγματεύσεις ένταξης έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο. Στα πλαίσια αυτών μπορούμε να πούμε ότι εκτιμούμε σε γενικές γραμμές την εκτίμηση του κυρίου Σφόποτα όπως παρουσιάζεται στην εκθεσή του. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πούμε δύο λόγια όσον αφορά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά από τα 35 10 κεφάλαια. Και βέβαια τα δέκα αυτά κεφάλαια είναι τα πιο δύσκολα που πρέπει να αντιπωστούν. Και έγιναν κάποια σχόλια ήδη όσον αφορά τα βασικά δικαιώματα, το δικαστικό, την καταπολέμηση της ε, διαφοράς, το ICT. Η Κομισιόν δεν δίνει η ημερομηνία για την ενδεχόμενη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή λέμε ότι έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο χωρίς να λέμε μέχρι πότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Όσον αφορά το γνωστό κεφάλαιο 23, δικαστικό και βασικά δικαιώματα των πολιτών, θα κάνουμε πραγματικά μια απογραφή της περαιτέρω προόδου της Κροατίας το Μάρτι και από εκεί και πέρα θα έχουμε ε, ενδεχομένω μια καλύτερη ιδέα πόσο γλίγορα μπορεί να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις. Τελευταία παρατήρηση. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες για να υποστηρίξει την Κροατία για να μπορέσει να πληρώσει τα ανοιχτά benchmark που υπάρχουν ακόμα. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά για εκείνους. Ε, υπάρχουν τα θέματα που πρέπει να λύσουν εκείνοι, τα σύνορα κλπ και να πρέπει να φτάσουν στα benchmarks. Ευχαριστώ. Πρώτα σε ευχαριστώ, Δόκτωρ Λάγκε. Ναι, ναι, ναι, θα, θα σας δώσω το λόγο, κύριε Σιγητά, για την τελική απάντηση, προφανώς. Θα σας ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Σφόβοτα. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομο Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια και την υποστήριξη της έκθεσης μου που υπάρχει και είναι αυτό και ένα θετικό μήνυμα προς την Κροατία. Αναφέρθηκαν διάφορα σημεία, παράγραφος 6, 8 κλπ. Και θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα αρχίσουμε εκεί με τα θετικά στοιχεία να τονίσουμε τι έχει ήδη καταφέρει να πετύχει η κυβέρνηση και μετά να προσθέσουμε την κριτική. Θα βρούμε οπωσδήποτε μια συνετική λύση και βρίσκω πολύ καλό που έχουμε πολλά κοινά σημεία και μπορούμε να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα θετικό για να βοηθήσουμε την Κροατία να λύσει τα τελευταία ανοιχτά θέματα. Και θα ήθελα να τονίσω ότι όταν εμείς δράσουμε ως κοινοβούλιο θα δράσουμε, αλλά τώρα η Κροατία θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Πρώτα, σε ευχαριστώ τον εισηγητή, κύριε Σουάβοντα. Δύο πληροφορίες με Σήμερα για τελευταία στιγμή εξετάσαμε το σύνολο της έκθεσης. 12 το μεσημέρι στις 14 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Θα ψηφιστεί <clears throat> στις 6 Ιανουαρίου στην Επιτροπή. Και η τελική ψηφοφορία προβλέπεται το Φεβρουάριο. Θα διακόψουμε τώρα. Στις 3 θα ξανασυζητήσουμε με την ανταλλαγή του Υπουργού Εξωτερικών και Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης του Βελγίου σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.